Dear colleagues, uh, we're going to make a start uh, with some announcements. Um, before we begin with the adoption of the agenda... Οι συνάδελφοι, ξεκινήσουμε με κάποιες ανακοινώσεις. Πριν περάσουμε στην ημερήσια διάταξη, θα διαβάσω μια δήλωση των διερμηνέων. Γνωρίζετε το ζήτημα για τους συναδέλφους που δεν το γνωρίζουν. Οι διερμηνείς σας ενημερώνουν ότι η εργασιακή διαμάχη λόγω των νέων όρων εργασίας ε, που επιβλήθηκαν μόνο μερός εξακολουθεί να ισχύει. Είμαστε στην τρίτη εβδομάδα. Οι διερμηνείς ε, έχουν κάνει πολλές ε, παραχωρήσεις. Η διοίκηση όμως δεν έχει κάνει καμία απόφυρα να έρθει σε επαφή μαζί μας για να επιλύσει την ε, σύγκρουση. Οπότε λένε οι διερμηνείς ότι ε, έχουν επιταχθεί και βεβαίω υπάρχει κάποια διακριτική μεταχείριση κάποιων γλώσσων γι' αυτό αποφάσισαν να μην κάνουν στάση εργασίας και δυστυχώς ε, μας ενημερώνουν ότι δεν θα υπάρξει καμία υπέρβαση του ωραρίου και η διερμηνία θα σταματήσει ακριβώς την ώρα που προβλέπετε. Σας ευχαριστώ λοιπόν για που ακούσετε αυτήν την ανακοίνωση. Ελπίζω να διάβασα καλά την ανακοίνωση, λέει Λοιπόν, έχουμε άρα αυτόν τον περιορισμό. Περνάμε τώρα στην έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Να προτείνω τις εξής αλλαγές. Το σημείο 5 θα είναι τώρα το σχέδιο ψηφίσματος για την ανθρωπιστική βοήθεια στις 11 η ώρα το 14 αφορά την συμφωνία με την Τινησία, όχι την Τουρκία. Ε, πρόκειτο περί τυπογραφικού λάθους. Το 33 είναι η παρουσίαση του σχεδίου έκθεσης για την αποστολή στην Βουλγαρία. Η κοινή επιχείρηση Frontex 12 με 14 Φεβρουαρίου αναβλήθηκε. Το 24 και 25 θα τα δούμε 15 λεπτά νωρίτερα και αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις εγκρίνει τη μυρίσια διάταξη. Για τα γλωσσικά ανέφερα βεβαίως το θέμα και επιπλέον δεν υπάρχει διερμηνία θα είναι διερμηνία σε όλες τις γλώσσες εκτός από κροατική, δανέζικη, μαλτέζικη και ιρλανδική περνάμε κατόπιν στην έγκριση των συστάσεων των συντονιστών ε, στο 205 έχουμε κάποιους εισηγητές που ορίστηκαν Πρώτα απ' όλα ο κύριος ε, Στέτινα του ΕΛΚΑ έχει οριστεί εισηγητής για την εφαρμοστική απόφαση του Συμβουλίου για την αυτόματη ανταλλαγή δεδομένων όσον αφορά την Κροατία. Ο κύριος Κρύπεκ του ECR εισηγητής για την εφαρμοστική απόφαση για τις ε, ψυχοτρόπες ουσίες. Ε, ένα θέμα από αυτές. Ο κύριος Κάρλος Κοέλιο του ΕΛΚΑ εισηγητής για τον κανονισμό για την ΒΙΖ και για τις νομοδοτήσεις η Άννα Γκόμεζ για την ε, νομοδότηση για το blockchain ο κ. Παύλ σοσιαλδημοκράτης δεν είναι των σοσιαλδημοκρατών λοιπόν εισηγητής ε, για την σύσταση μιας Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας. Μιχάλ Μπόνι, εισηγητής για την έκθεση Δίας Πρωτοβουλία για τη βιομηχανική πολιτική και την τεχνητή νοημοσύνη και τη ρομποτική. Εγκρίνονται οι συστάσεις αυτές των συντονιστών. Ωραία. Μετά. Πράξεις κατεφαρμογή και κατεξιοδότηση. Λάβαμε δύο σχέδια αποφάσεων. Ένα στις 11 Ιουνίου η Κομισιόν ε, ενέκρινε την εφαρμοστική οδηγία για συναγερμούς ε, και όπλα σημάτων ε, όσον αφορά τον έλεγχο οπλοκατοχής και στις 12 Ιουνίου ενέκρινε την εφαρμοστική οδηγία για την σήμανση πυροβόλων όπλων και των κύριων μερών τους. Επίσης για την εφαρμογή της οδηγίας για την οπλοκατοχή. Ε, το βασικό νομοθέτημα είναι η οδηγία 2017 κάθετος 853 που τροποποιεί την οδηγία του Συμβουλίου 91 κάθετος 477 ΕΟΚ για την ε, οπλοκατοχή. Σας είχαν ε, κοινοποιηθεί αυτά στις 15 ε, Ιουνίου, η ιστορική προθεσμία ε, ορίστηκε στις 25 Ιουνίου, εάν υπάρχει κάποια αντίρρηση και 26 Ιουνίου αντιστοίχω. οπότε ενημερώστε μέχρι τότε την γραμματεία αν υπάρχει κάποια αντίρρηση. Και μετά έχουμε μια ηλεκτρονική ψηφοφορία στις 11 και 4 σήμερα, οπότε να έχετε τις ε, κάρτες, της ψηφοφορίας Σε ποιον μιλάω, σε τέσσερις βουλευτές. Σας ευχαριστώ που ήρθατε. Οπότε, περνάμε τώρα στο σημείο 3, έκθεση του τριμερούς ε, διαλόγου και είναι μέρος της τακτικής ε, διαδικασίας του προϋπολογισμού. Είναι ανταλλαγή απόψεων για το σχέδιο προϋπολογισμού 2019, βιώτη για τις ε, ε, προτεραιότητες τη Επιτροπή μα. Ε, ο κύριος Βιώτη δεν είναι ο κύριο Χρυσόγονο. Ωραία. Λοιπόν, ο κύριος ε, Χρυσόγονο, λοιπόν, εισηγητής τη γνωμοδότηση τη Επιτροπή μα. Σα ευχαριστώ. Συγγνώμη, κύριε Χρυσόγονο. Ναι, ναι, έχετε το λόγο, ναι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σε μια κρίσιμη φάση όσον αφορά την εξέλιξη του ευρωπαϊκού εγχειρήματο. Η σωστή εφαρμογή των θεμάτων πολιτικών ελευθεριών, δικαιοσύνης και εσωτερικών είναι βασικό στοιχείο του ευρωπαϊκού εγχειρήματο. Μία περιοχή ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης είναι προαπαιτούμενο για την καταπολέμηση του εγκλήματος και να υπάρχει σωστή άσκηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων εντός της Ένωσης. Άρα το ύψο των οικονομικών πόρων που παρέχεται από το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο για το 2019 θα ε, είναι στο πλήρες ύψος του. Λόγω των ε, μεγάλων προκλήσεων, λόγω των αυξημένων αφήξεων μεταναστών στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει μεγάλη σημασία να δοθεί η απαραίτητη χρηματοδότηση έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασύλου να γίνει μια πλήρης η υπηρεσία η οποία θα σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα όλων των ετούντων. Στο πλαίσιο αυτό είναι επίσης σημαντικό η Frontex να έχει επαρκή χρηματοδότηση για να μπορεί να επιτελέσει την αποστολή της. Στο πλαίσιο αυτό, η πολύ σημαντική αύξηση των σχετικών ε, κονδυλίων ε, κατά 56% για να χρηματοδοτηθεί η νέα νομοθεσία του Δουβλίνου και ο φάκελος 175 εκατομμυρίων ευρώ που ζητήθηκε για την Ελλάδα θεωρούνται θετικά βήματα. Η κατάσταση στο τέλος του 2017 που κατέληξε στην ε, ανακατανομή 275 εκατομμυρίων ευρώ πιστώσεων πληρωμών από το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης ε, και Ένταξης λόγω ζητημάτων ικανότητας απορρόφησης κάποιων κρατών μελών πρέπει να μην επαναληφθεί στο μέλλον. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να υπάρξει μία γραμμή του προϋπολογισμού για κάθε έναν στόχο για να μπορέσει η Επιτροπή μας να παίξει τον ρόλο της ε, του ελέγχου και της διαφάνειας της κοινοτικής χρηματοδότησης όσον αφορά την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων πρέπει να τονίσουμε την ε, σημασία χρηματοδότησης ε, μηχανισμών εποπτείας σε ζητήματα δικαιοσύνης και εσωτερικών καθώς είναι προφανές ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα υφίστανται πιέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση προτείνουμε η προϋπολογισμοί της Υπηρεσίας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Θεμελιωδών Προσωπικών Δεδομένων να αυξηθούν και επίσης θα πρέπει η Ιουλίζα να έχει επαρκής πόρους το 2019 για να μπορεί να προσλάβει το προσωπικό και την έμπειρο γνωμοσύνη που χρειάζεται για να επιτελέσει τα καθήκοντά της παρά το ότι αυτό δεν συμβαίνει με την τωρινή πρόταση της ε, Κομισιόν στο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027. Όσον αφορά το Ταμείο Εσωτερικής Ασφαλείας, ε, πρέπει να τονίσουμε ότι η ενίσχυση της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του σοβαρού εγκλήματος, όπως και του κύβερνο εγκλήματος, είναι προτεραιότητες της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ. Ως εκ τούτου. Δεδομένου του σημαντικού της ρόλου στην καταπολέμηση διαφόρων μορφών εγκλήματος και τη συνεργασίας με τρίτες χώρες, η Europol θα έχει επαρκή χρηματοδότηση. Το ίδιο ισχύει και για την χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας. Επιπλέον, ε, η εφαρμογή της αναθεώρησης ε, του, της εντολής ε, του δικτύου για με συγχωρείτε, τις υπηρεσίες για την ασφάλεια των δικτύων θα πρέπει να ενισχυθεί για να καταπολεμήσουμε το κυβερνό έγκλημα. Επιπλέον, ο προϋπολογισμός της Eurojust του δικαστικού δικτύου θα πρέπει να ενισχυθεί για να υπάρξει ο κατάλληλος συντονισμός έρευνων και διώξεων μεταξύ των αρμοδίων αρχών των κρατών μελών. Όμως, η ουσιαστική μείωση στο πι 2021-2027 των πιστώσεων ε, υποχρεώσεων του προγράμματος δικαιοσύνης και της Eurojust είναι κάτι το αντιπαραγωγικό. Η μείωση αυτή είναι κάτι το οποίο δεν στέκει δεδομένη τη ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα και των πολιτικών προτεραιοτήτων και θα πρέπει να αναθεωρηθεί από την άλλη ο προπολογισμό 4,9 ε, εκατομμυρίων ευρώ για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι μια θετική καινοτομία στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών. Συμπερασματικά, πρέπει να έχουμε κατά νου ότι η σωστή εφαρμογή του προπολογισμού, ειδικά στον κρίσιμο τομέα πολιτικών ελευθεριών, δικαιοσύνης και εσωτερικών θα συνεχίσει να ενισχύει την εφαρμογή των θεμελιωδών αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως η προστασία ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλληλεγγύη, κοινή συνεργασία και δημοκρατία. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Ξόνα. Ένας σκιώδης ε, εισηγητής, ο κύριος Μάμικινς για τους σοσιαλδημοκράτες. Α, ο κύριος Βιώτη ήρθε, μάλιστα. Ναι, ναι, μετά τον κύριο Μάμικινς θα σας ακούσουμε. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα είμαι σύντομο. Θέλω να τονίσω τρία σημαντικά θέματα για τον προπολογισμό τη επόμενη χρονιά. Είναι τα δικονομικά δικαιώματα όλων των ετούντων που βρίσκονται σε ε, κέντρα υποδοχής και όλα τα ζητήματα της υποστήριξης της μετανάστευσης. Δεύτερον, θα πρέπει η Επιτροπή Θεμελιωδών Ελευθεριών να μπορέσει να παίξει το ρόλο της για να ασκήσει τον κοινοβουλευτικό έλεγχο της χρηματοδότησης στην Ένωση και τρίτον θα πρέπει να ε, ενισχύσουμε το EDPS το, και το, την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ε, την, την αρχή ε, προστασία των προσωπικών δεδομένων. υπήρξαν κάποιες ε, τροπολογίες τις οποίες έχω επισημάνει σε συγκεκριμένες παραγράφους τις οποίες δεν θα αναφέρω τώρα αλλά είναι πολύ σημαντικές και τις έχουμε συζητήσει με τον εισηγητή. Σας ευχαριστούμε κύριε Μάπικινς. Ο κύριος Βιώτη που είναι ο εισηγητής για τον ε, προπολογισμό. Κύριε Χρυσόγονα θα θέλετε να πάρετε το λόγο με... Όχι ευχαριστώ λέει ο κύριος Χρυσόγωνος. Θα σας δώσω μετά το λόγο για τα συμπεράσματα. Κύριε Βιώτη, λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς, να ζητήσω συγγνώμη για την καθυστέρηση. Ζητώ συγγνώμη, λοιπόν, για την καθυστέρηση. Οφείλεται στη γνωστή κίνηση των Βρυξελών και ζητώ συγγνώμη και με από την μέλη της Επιτροπής και σας ευχαριστώ που με προσκαλέσατε σε αυτή την ε, συζήτηση. Εγώ έχω κάνει ένα γύρο όλων των επιτροπών ήδη και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα να μπορέσω να συζητήσω με τους συναδέλφους ε, ιδιαίτερα στις ε, εξειδικευμένες επιτροπές διότι ε, ναι μεν ε, ε, γνωρίζω τι γίνεται στην Επιτροπή Προπολογισμών, αλλά τις λεπτομέρειες τις γνωρίζω επιφανειακά. Ευχαριστώ πολύ για την επιστολή που μου στείλατε. Τα ξέρετε τα θέματα, δεν χρειάζεται να τα επαναλάβω εγώ. Μου τα έγραψε το Μάρτιο ο Πρόεδρος. Υπάρχουν όμως κάποια πράγματα στα οποία θα ήθελα να σταθώ και θεωρώ ότι είναι απαραίτητο να επενδύσουμε ε, ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως επισημαίνετε και εσείς. Στον τομέα του ασύλου και της μετανάστευσης βεβαίως η χρηματοδότηση πρέπει να είναι παρκές για την αλλαγή της ΕΑΣΟ ε, και να γίνει ε, μια διαφορετική υπηρεσία που έχει συγκεκριμένο στόχο, τον οποίο συμμερίζομαι, αλλά είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί, όχι τόσο από οικονομική σκοπιά, όσον αφορά τη διαμόρφωση του προπολογισμού. Δηλαδή, τον ε, επιμερισμό του ΆΜΙΦ σε τέσσερις ε, γραμμές προπολογισμού, όπως επίσης και γραμμές προϋπολογισμού οι οποίες θα είναι πολύ καλά σταθμισμένες και θα αφορούν ε, τα θέματα έρευνας και διάσωσης στη θάλασσα. Πρόκειται για επιχειρήσεις τις οποίες επικροτώ και θα προσπαθήσουμε να συμπεριλάβουμε στη συζήτηση ε, στην ε, διαδικασία της συνδιαλλαγής. Αλλά πιστεύω ότι θα πρέπει να προετοιμαστούμε πάρα πολύ, ιδιαίτερα για το επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, στο οποίο δεν θα επισέλθω βέβαια τώρα, όταν θα υπάρξει το νέο πλαίσιο. Τώρα, όσον αφορά τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων, σίγουρα πρέπει να υπάρχει επαρκή ε, χρηματοδότηση για το Frontex, καθώ επίση και πόροι και προσωπικό για το EU Lisa, γιατί θα αναλάβει και νέα καθήκοντα. αυτό ήμασταν απόλυτα σαφεί και ω Επιτροπή Προπολογισμών, αλλά και ω Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκό Πάντα ζητάμε από τα κράτη-μέλη, διότι γνωρίζετε ότι ούτω ή άλλω με αυτού ε, θα διαπραγματευτούμε. Για κάθε νέα ανάγκη χρειάζεται νέο φρέσκο χρήμα. Οποιοδήποτε νέο καθήκον ανατίθεται πρέπει να σημαίνει και νέα κονδύλια και νέο προσωπικό. Δεν μπορεί οι υπηρεσίε και οι οργανισμοί να κάνουν τη δουλειά ε, που κάνουν συν επιπλέον πράγματα με λιγότερο προσωπικό ε, από όσο χρειάζεται. Όσον αφορά την εσωτερική ασφάλεια και την ε, δικαστική και αστυνομική συνεργασία, δεδομένου ότι υπάρχουν τα συνοριακά θέματα, η διακίνηση ανθρώπων κλπ. Πρέπει να υπάρχει επαρκή χρηματοδότηση για οργανισμούς όπως η Eurojust, τη Νέα Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και τη Europol. Επίσης, πάντα στον τομέα της μετανάστευση και του ασύλου υπάρχει ε, χρηματοδότηση για την αντικατάσταση των, ε, ε, του, μέσου για την ανθρωπιστική βοήθεια που θα μπορούσε να δημιουργήσει προβλήματα στη διαδικασία της συνδιαλλαγής. Αναφέρθηκε μεγαλύτερη πρικοδότηση για την υπεδοχή και ένταξη ετούντων άσυλο. Για την ΕΑΣΟ είπαμε έλεγχος και διαχείριση των συνόρων και να μπορέσουμε να έχουμε κατάλληλη πρικοδότηση και ανθρώπινους πόρους για το Ιουλίσα. Για τους πόρους των υπηρεσιών και των οργανισμών, ε, το τελευταίο το οποίο θα πω σε αυτή τη σύντομη παρουσίαση. Θα θυμάστε ότι πέρσι καταφέραμε στη διαδικασία της συνδιαλλαγής να κάνουμε κάτι το οποίο δεν ήταν εμένα αυτό το οποίο επιθυμούσαμε στο σύνολό του, αλλά θέλαμε για τη Europol, την EASO και τη Eurojust να έχουμε μια μικρή αύξηση και κονδυλίων και προσωπικού. Ο στόχος φέτος είναι και πάλι να συνεχίσουμε προς αυτή την ε, κατεύθυνση, με εξαίρεση βεβαίω το γεγονό ότι το Συμβούλιο θα ζητήσει κατά πάσα πιθανότητα για άλλε υπηρεσίε και για άλλα κονδύλια μειώση του προσωπικού και τη χρηματοδότηση. Και εδώ θα ήθελα επίσης να είμαι σαφής. Εάν δεν υπάρξει αύξηση πόρων από πλευράς ε, Συμβουλίου, δεν υπάρξει δηλαδή κατάλληλη απάντηση, εμείς ε, κατά πάσα πιθανότητα θα επιμείνουμε και υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να μην υπάρχει κανένα αποθεματικό για αύξηση χρηματοδότησης, για πιλωτικά προγράμματα και προπαρασκευαστικές δράσεις. Και σε αυτό πρέπει να είμαστε σαφείς. Μια τελευταία παρατήρηση που είναι περισσότερο πολιτικής φύσεως παρά τεχνικής, είναι ότι όπως γνωρίζετε και θα φαντάζεστε, εμείς θα δεχτούμε τα περισσότερα από τα αιτήματα που θα μας ε, κάνει, μας κάνει ήδη η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ αλλά πρέπει να υπάρξει μια νέα συμφωνία κυρίων με το ε, Συμβούλιο. Διότι αν το Συμβούλιο, το οποίο από ό,τι φαίνεται, δεν θέλω βέβαια εδώ να μιλήσω για μονομενα περιστατικά, αλλά δεδομένω και τη νέα κυβέρνηση στην Ιταλία, δεδομένου και του προσανατολισμού που φαίνεται να ακολουθεί το Συμβούλιο. Αν το Συμβούλιο σκοπεύει να στοχεύσει πολύ περισσότερο στη διαχείριση της μετανάστευσης, στη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών κλπ. πρέπει να υπάρχουν κατάλληλοι πόροι. Δεν μπορεί να ζητάμε από το Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αντιμετωπίσουν νέες ε, ε, προκλήσεις, νέες αποστολές, νέα προγράμματα και νέα καθήκοντα χωρίς να υπάρχει κατάλληλη χρηματοδότηση και γι' αυτά αυτό πρέπει να αποτελέσει και κόκκινη γραμμή για μας, ε, πρέπει να αποτελέσει κόκκινη γραμμή για όλο το κοινοβούλιο θεωρώ, διότι ε, η Δάλος Δεν μ' αρέσει να χρησιμοποιώ βεβαίω αυτόν τον όρο, αλλά η Δάλος όχι μόνο θα γίνουμε λαϊκιστικές δυνάμει, αλλά θα γίνουμε απλώ και δι... λαϊκιστικέ και οργανώσει λαϊκιστικέ, διότι ζητάμε να εφαρμοστούν πολιτικέ χωρί να διαθέτουμε και τα κατάλληλα κονδύλια. Ο στόχος μου λοιπόν και ε, η μέθοδος που θέλω να ακολουθήσω είναι να υπάρχει η μέγιστη δυνατή αποδοχή, ο μέγιστος δυνατός αριθμός συναδέλφων που θα εγκρίνουν την ε, ε, εντολή για την ε, διαπραγμάτευση στον τριμερή διάλογο, διότι αυτό είναι και το ισχυρό χαρτί για τον εισηγητή για τον προπολογισμό και αυτό είναι σημαντικό όχι μόνο από πλευράς πολιτικών ομάδων, αλλά πλήρης υποστήριξη από κάθε επιτροπή. Και νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Thank you very much, Daniel. <clears throat> Thank you. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Ήταν ξεκάθαρη τοποθέτησή σας. Ακολουθούμε λίγο περίεργη διαδικασία γιατί κάθε συνάδελφος έχει έρθει σε διαφορετική χρονική στιγμή. Αν κάποιος άλλος από τους σκιώδες θα ήθελε το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όταν συζητούσαμε το περιεχόμενο της επιστολής που θα στείλει η Επιτροπή Λίμπε στον πρόεδρο της Επιτροπής Προϋπολογισμού, είχα πει ξεκάθαρα ότι πρέπει να είναι σαφείς οι προτεραιότητες μας. Και πιστεύω ότι στον τομέα της δικαιοσύνης και των ιστορικών υποθέσεων θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι εκείνα τα κράτη-μέλη που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή και πρέπει να αντιμετωπίσουν τους ετούντε άσυλο θα έχουν την υποστήριξη που χρειάζονται από το, ε, την ΕΑΣΟ και από τη Frontex. Γνωρίζω ότι έχουμε νέες νομοθετικές, νέα νομοθετήματα και εργαλεία. Όμως εγώ θα ήθελα να ε, δω αυτό να συμβαίνει ως αποτέλεσμα της συνήθους διαδικασίας του μέρους διαλόγου. Θα πρέπει επίσης να έχουμε τους κατάλληλους πόρους για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και του λαθρεμπορίου. Γνωρίζουμε ότι οι χώρε που βρίσκονται στα εξωτερικά σύνορα τη Ένωση αισθάνονται ότι δεν έχουν την απαιτούμενη υποστήριξη. Θα πρέπει να δοθούν οι απαιτούμενοι πόροι και στον τομέα του ασύλου. Πιστεύω ότι περισσότεροι πόροι θα πρέπει να δοθούν στη Frontex, έτσι ώστε να παράσχει βοήθεια ε, στα κράτη-μέλη με τον έλεγχο των εξωτερικών του συνόρων. Επίση, πιστεύω ότι πρέπει να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες ε, ευελιξίας ε, έτσι ώστε να εφαρμόσουμε τις ε, πολιτικές ε, με επιπλέον πόρους. Με βάση τις προτάσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμού παρά το γεγονό ότι αναγνωρίζονται ότι ο τομέας της ασφάλειας είναι σημαντικός, δεν, δεν έχει δοθεί αντίστοιχη ε, έμφαση στα ζητήματα της μετανάστευση. τα προβλήματα της μετανάστευση μπορούν να απεσταθεροποιήσουν όχι μόνο κάποια κρατημέλη, αλλά ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να λύσουμε το πρόβλημα της παράτυπης μετανάστευσης, γιατί διαφορετικά θα έχουμε ε, τεράστια προβλήματα που δεν θα μας επιτρέψουν να σκεφτούμε άλλες προτεραιότητες όπως για παράδειγμα την καινοτομία. Στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το νέο Πουδουπού το συνολικό ε, ποσό για την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών και την έλεγχο των εξωτερικών συνόρων έχει τριπλασιαστεί μέχρι 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Ε, θα πρέπει να τονίσουμε την, επίσης τη σημασία που έχει η οικονομική υποστήριξη των προγραμμάτων για την καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης, την ε, διαχείριση κρίσεων και την κυβερνοασφάλεια. Όσον αφορά τώρα τον προπολογισμό για το εσωτερικό, την εσωτερική ασφάλεια, θα πρέπει να ε, ε, ενισχυθούν οι πόροι για την αστυνομική και δικαστική συνεργασία. Θα πρέπει να δοθούν κατάλληλοι πόροι στην λύσα, περίπου 100 εκατομμύρια ευρώ, Μιας και από το 2019 η Ιουλίσσα θα κληθεί να παίξει πολύ σημαντικότερο ρόλο, θα πρέπει να έχει στη διάθεσή τη του πόρου που χρειάζεται. Είναι περιορισμένοι οι πόροι που έχουμε στη διάθεσή μα για να πετύχουμε όλου του στόχου πολιτική για τα επόμενα δύο χρόνια που θα πρέπει να καλύψουμε με το τρέχον πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Επομένω, θα πρέπει να φροντίσουμε να του αξιοποιήσουμε αποτελεσματικά και να τους αποδώσουμε στους πόρου, τους πόρους εκείνους στα προβλήματα που επηρεάζουν άμεσα το μέλλον της Ευρώπης όπως η μετανάστευση. Προσβλέπω στη συζήτηση που θα έχουμε για τον προπολογισμό του 2019 έτσι ώστε να τονίσουμε για άλλη μια φορά ποιες είναι οι προτεραιότητές μας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Πράγματι τα θέματα αυτά θα πρέπει να τα συζητήσουμε περαιτέρω και είμαι σίγουρος ότι και ο συζητής θα ήθελε να απαντήσει, αλλά θα πρέπει να διακόψουμε αυτή τη συζήτηση εδώ γιατί έχει έρθει ο Υπουργό ε, Μεταναστευτική Πολιτική τη Ελλάδα και ο χρόνο μα πιέζει. Σας ευχαριστώ κύριε Βιώτη για την παρέμβασή σας. Ευχαριστώ και τον εισηγητή τον κύριο Χρυσόγωνο, ευχαριστώ και τους ε, σκιώδεις εισηγητές. Έχει έρθει ο Έλληνας Υπουργός, μπορούμε να τον καλέσουμε.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 Colleagues, we can move now to point... Ωραία, συνάδελφοι, μπορούμε να συνεχίσουμε με το σημείο 4 της τη διάταξη. Θα ήθελα να καλωσορίσω τον κύριο Δημήτρη Βίτσα, Έλληνα Υπουργό μεταναστευτική πολιτική. Είναι ένα θέμα πολύ σημαντικό. Σε κάθε περίπτωση θα θέλαμε να συζητήσουμε με τον νέο Υπουργό. Το ζήτημα όμω είναι ακόμα μεγαλύτερο, ακόμα σημαντικότερο. Σήμερα είναι και η Παγκόσμια Μέρα για του πρόσφυγε. Θα ήθελα να σα καλωσορίσω Γνωρίζω ότι πολλοί από του συναδέλφου γνωρίζουν ήδη τον Υπουργό από προηγούμενε συναντήσει και συζητήσει. Εχθέ ε, κάναμε μια συζήτηση για το θέμα και γνωρίζω ότι οι συνάδελφοι θα ήθελαν να ακούσουν από τον Υπουργό αυτό που λέμε το μακροπρόθεσμο επίπεδο, τι συμβαίνει και ποια είναι τα τρέχοντα προβλήματα, καθώ επίση για το τι πρόκειται να γίνει, τι φαντάζεστε ότι μπορεί να γίνει στην επόμενη συνάντηση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου την επόμενη εβδομάδα, καθώς επίσης και τα ζητήματα που σας απασχολούν στην ε, Ελλάδα, στην Αθήνα. Οι συνάδελφοι εδώ ε, είναι γνώστες του θέματος και θέλουν να έχουν μια ουσιαστική συζήτηση μαζί σας. Δεν θέλω να μακρηγορήσω, θέλω να σας δώσω αμέσως το λόγο για να έχουμε χρόνο μετά ε, και τη δυνατότητα να συζητήσουμε με τους συναδέλφους. Έχετε φέρει ένα βίντεο ε, και επί τη ευκαιρία της Παγκόσμιας ημέρας προσφύγων και νομίζω μπορούμε να το δούμε. Μπορούμε. Έρχεται το βίντεο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 Sir, if you could um, warm welcome again and please go ahead and we'll... Καλώς ορίσατε και πάλι κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο μας. Σας ευχαριστώ πολύ, θα μιλήσω ελληνικά. Consular and uh, will be, I think, enough to inform you what is happening in Europe and in uh, Greece uh, right και θα σας ενημερώσω για το αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα και στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Χαρά και τιμή για μένα σήμερα που τιμάμε την Παγκόσμια ημέρα του πρόσφυγα που μου δίνετε την ευκαιρία να απευθυνθώ στην Επιτροπή σας και μέσα αυτού να καλημερίσω και τα αξιότιμα μέλη της Επιτροπής. Ο ρόλος που διαδραματίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο σχεδιασμό της διαχείρισης της μεταναστευτικής και προσφυγικής κρίσης και στη χάραξη μιας πανευρωπαϊκής πολιτικής στους τομείς του ασύλου και της μετανάστευσης είναι κέριος και επίκαιρος όσο ποτέ άλλοτε. Μια πολιτική με σεβασμό στις κοινέ ευρωπαϊκές αξίες, με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, στη βάση των ευρωπαϊκών συνθήκων και των κανόνων του διεθνούς δικαίου. Επιτρέψτε μου να επικεντρωθώ σε ορισμένα σημεία του ζητήματος όπως εμφανίζεται σήμερα, και να πω τη γνώμη μου σχετικά με τις εξελίξεις για των συζητήσεων για τον κανονισμό για το Δουβλίνο 4 και για την κατάσταση στην Ελλάδα, πώς διαχειριζόμαστε, ποιο είναι το πρόγραμμά μας το δεύτερο εξάμεινο του 2018 και το 2019. Αλλά πριν αναφερθώ σε αυτά, ε, θέλω να μοιραστώ μαζί σας μια βασική σκέψη. Η κοινή ευρωπαϊκή μας πορεία, η Ευρωπαϊκή Ένωση, αναζητεί και απαιτεί συνεχή διάλογο, βλέμμα στραμμένο στο μέλλον και βέβαια συμβιβασμούς. Όμως όλα τα, τα παραπάνω πρέπει να γίνονται σε μια κοινά παραδεκτή βάση, αλλιώς γυρνάμε στην αρχή, όταν δεν υπήρχε Ευρωπαϊκή Ένωση. Χωρίς κοινέ αξίες, χωρίς κοινού κανόνες, χωρίς κοινέ ε, συνθήκες. Και εδώ είναι το ζήτημα και το ερώτημα της εποχής που αφορά και το προσφυγικό ή αφορά κατά κύριο λόγο το προσφυγικό. Η συνθήκη της Γενέβης, το πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης και όσες συνθήκες και συμφωνίες πηγάζουν από αυτή, ισχύουν, ναι ή όχι. Όταν μιλάμε για αλληλεγγύη, μιλάμε για αλληλεγγύη προς ανθρώπους και συνακόλουθα για αλληλεγγύη συνεργασία μεταξύ των κοινωνιών και των κρατών για να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους ή μιλάμε για αλληλεγγύη μεταξύ κρατών για να αποτρέψουμε την ευθύνη διαχείριση του ζητήματος. Η απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα είναι οδηγός και όλα τα επιμέρους μέτρα, συμφωνίες κτλ. κρίνονται πλέον από αυτή την απάντηση και κρίνονται και τα πρακτικά μέτρα. Είναι εμφανές ότι η δικιά μου άποψη είναι στο πρώτο κομμάτι του ερωτήματος. Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε σαν Ευρώπη στους τομείς της μετανάστευσης και του ασύλου απαιτούν συνεργασία ανάμεσα σε όλους τους εμπλεκόμενους στη βάση των κοινών μας αξιών, του διεθνούς δικαίου και των αρχών της αλληλεγγύης και του επιμερισμού των ευθυνών. Απέχουμε πολύ από το στόχο αυτό, καθώς δεν αντιλαμβάνονται όλες οι χώρες της Ευρώπης και όλες οι ευρωπαϊκές πολιτικές δυνάμεις με τον ίδιο τρόπο τα πράγματα. Ποιος είναι αυτός ο στόχος? Τίποτα λιγότερο από μια θεσμοθετημένη ευρωπαϊκή πολιτική για τη μετανάστευση και το άσυλο, που θα περιλαμβάνει οπωσδήποτε τους εξής άξονες. Πρώτο, νόμιμες και ασφαλείς οδούς για τους πρόσφυγες, ώστε να μην στρέφονται στα κυκλώματα διακίνησης. Δεύτερο, δίκαιο και βιώσιο κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου, που να είναι ανθεκτικό σε κρίσεις και δεν θα επιβαρύνει αποκλειστικά και μόνο τα κράτη-μέλη στα εξωτερικά σύνορα και τρίτο, ενίσχυση της συνεργασίας με τις τρίτες χώρες για να αντιμετωπίσουμε τις γενεσιουργές αιτίες της μετανάστευσης. Ως τώρα, και για να, μην, μιλάμε την γλώσσα της αλήθειας, οι εξελίξεις στον ευρω... ευρύτερο ευρωπαϊκό περίγυρο δεν είναι θετικές. Οι πόλεμοι και οι σειράξει συνεχίζονται και δυστυχώς δεν προβλέπεται να τερματιστούν σύντομα. Οι κοινωνικές ανισότητες αυξάνονται και μας προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία οι επιδεινούμενες συνθήκες διαβίωσης των προσφύγων και των εκτοπισμένων στο Λίβανο, την Ιορδανία, το Ιράκ, τη Συρία και την Τουρκία, σύμφωνα και με τις πρόσφατες εκθέσεις της ΥΠΑ της και του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης. Οι απαντήσεις σε αυτές τις προκλήσεις βρίσκονται στη συνεργασία, στη συνεργασία όλων μας. Η Ευρώπη θα πρέπει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Η επαναγκατάσταση θα πρέπει να είναι το κύριο εργαλείο για τη διαχείριση των ροών. Ένα γενναιόδωρο και φιλόδοξο πρόγραμμα επανεγκατάστασης θα αδρανοποιήσει τα κυκλώματα των διακινητών, θα δώσει δυνατότητα σε όσους δικαιούνται να έρθουν νόμιμα και με ευταξία στην Ευρώπη. θα πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειές μας και να είμαστε αμήλικτοι προς τα κυκλώματα των διακινητών που εκμεταλλεύονται την ανθρώπινη απελπισία. Ένα από τα πιο κύρια ζητήματα είναι σήμερα αυτό της αναθεώρησης του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου και ειδικότερα του κανονισμού του Δουβλίνου. Θέλω να είμαι καθαρός. Η Ελλάδα υποστηρίζει την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού, της Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Βρισκόμαστε σχεδόν ταυτόσιμοι σε αυτές τις ε, θέσεις και με χαρά υποδεχθήκαμε την τελευταία επιστολή του κυρίου Ταβιάννη προς τον ε, Έλληνα Πρωθυπουργό και ελπίζουμε ότι και οι άλλοι ηγέτες των κρατών μελών να την υποδεχθούν με τον ίδιο ε, τρόπο. αυτό είναι θα λέγαμε το επιθυμητό. Αυτό θα λέγαμε το είναι το επιθυμητό. Αυτό δηλαδή που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει καταλήξει. Συγχρόνως όμως ξέρουμε ότι στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τα πράγματα δεν είναι έτσι. Τα πράγματα πολλές φορές πηγαίνουν προς μια κατάσταση όπου δεν βρίσκεται λύση. Η θέση της Ελλάδας είναι ότι συμπαρίσταται στην προσπάθεια που κάνει η Βουλγαρική Προεδρία να βρεθεί ένας ανεκτός συμβιβασμός, προοδευτικός συμβιβασμός. Γι αυτό, το, γι' αυτό το λόγο θεωρούμε ως βάση για συζήτηση, παρά το γεγονός ότι έχουμε πολλές διαφορετικές ε, γνώμες, το κείμενο της Βουλγαρικής ε, Προεδρίας. Και εναντιονόμαστε σε, αυτούς, σε αυτά τα κράτη-μέλη που λένε ότι αυτό πρέπει να πάρθει ολόκληρο πίσω και να ξεκινήσουμε μια συζήτηση από την αρχή. Ένα δεύτερο ζήτημα που με επιμονή βάζουμε είναι ότι και εδώ πέρα χρειάζεται μια πίεση από τη μεριά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, ακόμα μεγαλύτερη από αυτή που κάνει ότι είναι καιρός γρήγορα να αρχίσει η διαδικασία των τριλόγων ώστε να βρεθεί μια τέτοια ε, κοινή λύση. Και τέλος, θεωρούμε ότι όπως ήρθαν τα 7 νομοθετήματα μαζί, ως πακέτο θα πρέπει να αντιμετωπιστούν και με αυτή την λογική εμείς ε, θεωρούμε ότι δεν πρέπει να σπάσουν σε μια διαδικασία στο επόμενο ε, διάστημα. Σαν πέντε χώρες ε, μέλη που είναι χώρες πρώτης υποδοχής προσπαθήσαμε από κοινού να παρέμβουμε σε αυτή τη συζήτηση και διατυπώσαμε 13 θέσεις ε, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Τέσσερις από αυτές έγιναν δεκτές. Εννέα δεν έγιναν δεκτές. Βέβαια όλα αυτά έχουν συμβεί εδώ και δύο περίπου ε, μήνες. Από τότε έχουν γίνει εκλογές, έχουν, έχει αλλάξει κάπως το ε, κλίμα, αλλά θεωρούμε ότι αυτές οι 13 θέσεις, οι οποίες είναι αντίστοιχες με τις αντίστοιχες θέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα πρέπει να γίνουν αποδεκτές. Παρόλα αυτά, δεχόμαστε να μπούμε σε μια τέτοια συζήτηση, ακριβώς για να βρούμε ε, λύση. Αλλά πρέπει να γίνουν αποδεκτές μια σειρά θέσεις που προβάλλουν οι χώρες της πρώτης υποδοχής, γιατί αυτές κατά κύριο λόγο σηκώνουν το κύριο ε, βάρος. Για μας, επαναλαμβάνω, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να υπάρχει επιμερισμός και όχι περαιτέρω επιβάρυνση του υποποίηση ήδη κράτου μέλους πρώτης υποδοχής με πρόσθετες υποχρεώσεις, περίπλοκες διαδικασίες που δεν πρόκειται να τηρηθούν, δεν μπορούν να τηρηθούν, όσο και αν ε, ενισχυθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες του. Δεν είναι λογική ότι δίνουμε σε κάποια κράτη-μέλη χρήματα και αυτές ας αναλάβουν το βάρος. Πρέπει όλο το βάρος να επιμεριστεί και η Ευρώπη είναι ικανή να το αντέξει. Και σε αυτό πρέπει να συμβάλλουν και είναι καλές οι ιδέες που έχουμε μελετήσει του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όλα τα κράτη-μέλη, ακόμα και υπό την πίεση κάποιας ε, ποινής. Θα ήθελα να αναφερθώ αν αυτές είναι οι καταρχήν οι θέση μας όσο αφορά το Δουβλίνο, ε, στην κατάσταση όπως είναι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Είδατε το βίντεο. Δεν είμαστε στο 2015. Και επειδή μια, γίνεται μια συζήτηση στην Ευρώπη δεν πρόκειται να επανέλθουμε στο 2015 γιατί δεν υπάρχουν τα αντικειμενικά στοιχεία να γυρίσουμε στο το 2015. Γιατί η συζήτηση στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή αντί να γίνεται για την ανακατανομή γίνεται λες και αύριο το πρωί θα έχουμε επανάληψη του 2015. Και αυτό θα πρέπει να απορριφθεί γιατί μας βάζει σε μια άλλη ατζέντα. Αυτό είναι το ε, βασικό ζήτημα. Αντιμετωπίσαμε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης, συνεχίζουμε την προσπάθειά μας. Τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά σε σχέση με το 2015, χωρίς να λέω ότι δεν υπάρχουν δυσκολίες και αδυναμίες. Αλλά από εκείνη την κατάσταση μέχρι τα τώρα είμαστε έτη φωτός ε, μπροστά. Σήμερα, χωρίς να παρουσιάσω μια εξοραϊσμένη εικόνα, η εικόνα είναι ως εξής. Στην Ελλάδα υπάρχουν 60.000 πρόσφυγες και μετανάστες. Από αυτούς περίπου 16.000 είναι στα νησιά. Υπήρξε μια αύξηση των ροών από την Τουρκία στο δεύτερο εξάμεινο του 2017 και το πρώτο τετράμινο του 2018. Δεν θα μπω στους συγκεκριμένους αριθμούς, η αύξηση όμως ήταν μεγάλη ιδιαίτερα τον Απρίλιο στα ε, χερσαία μας σύνορα. Αυτό δημιούργησε μια ασφιχτική κατάσταση στο ελληνικό σύστημα υποδοχής και ασύλου, ιδιαίτερα στα νησιά του ε, Αιγαίου αλλά και στον Εύρο. Είχαμε μια συνεχή επαφή με την Κομισιόν, τον κύριο Αβραμόπουλο και την Βουλγαρική Προεδρία. Είχαμε μια συνεργασία με την τουρκική πλευρά. Έγιναν δύο συναντήσεις σε υψηλό τεχνικό επίπεδο στην Κωνσταντινούπολη και στην Αθήνα αποτέλεσμα αυτών των συναντήσεων, βασικό αποτέλεσμα ήταν ότι επανήλθαν οι ροές στο επίπεδο του Μαΐου του 2017, δηλαδή πολύ πιο ε, χαμηλές. 6.600 πρόσφυγες ε, μπήκαν στην Ελλάδα τον Απρίλιο, 3.500 τον Μάιο και 1.500 τον ε, Ιούνιο. Καταλαβαίνετε, όσοι 15 του Ιουνίου. Καταλαβαίνετε την ε, διαφορά. Πρόθεση και βούληση της ελληνικής πλευράς είναι η ειλικρινή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με την Τουρκία για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ε, ροών. Επειδή τελευταία δημιουργείται μια αφήγηση, μια ιστορία για την ε, λεγόμενη Αδριατική Οδό των Δυτικών Βαλκανίων, επιτρέψτε μου να υπογραμμίσω ότι όσο και αν ε, αναζητούμε δεν υπάρχουν στοιχεία από αυτούς που τη λένε. Και όσο αφορά ε, εμάς, δεν υπάρχουν δευτερογενείς ροές από την Ελλάδα προς τις γειτονικές χώρες και προς χώρες της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης. Άρα προκαλούμε και προσκαλούμε να αναδειχθούν στοιχεία, γιατί τα στοιχεία που έχουμε εμείς λένε ότι από την Αλβανία όλο το 2017 έγιναν 18 αιτήσει επανεισδοχή στην Ελλάδα και ως σήμερα το 2018 έγιναν τρεις, τρεις, αριθμός τρεις μόνο αιτήσει επανεισδοχής. Αυτή τη στιγμή η πρώτη και κύρια έγνοια μας είναι η όσο δυνατόν άμεση αποσυμφόρηση των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου ιδιαίτερα της Λέσβου και της Σάμου, που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών, λόγω της γεωγραφικούς τους, της θέσης στα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης. Ο υπερπληθυσμό σε αυτά τα δύο κάμπ ε, δημιουργούν προβλήματα και στις συνθήκες διαβίωσης των προσφύγων, προσφύγων και των μεταναστών, όσο και στι τοπικέ κοινωνίε των νησιών αυτών. Ή για να διορθώσω. Δεν υπάρχουν πρόσφυγες και μετανάστες, κατά κύριο λόγο για τις υπηρεσίες ασύλου. Υπάρχουν ετούντες άσυλο, ετούντες διεθνούς προστασίας. Και όσοι έρχονται στην Ελλάδα κάνουν τέτοιου είδους αίτηση. Αυτό πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας. Το πρώτο λοιπόν ζήτημα είναι η επιτάχυση των διαδικασιών ασύλου με πλήρη σεβασμό στα δικαιώματα των ετούντων. Υιοθετήσαμε στα μέσα Μαΐου ένα νέο νόμο για το άσυλο η φιλοσοφία αυτού του νέου νόμου βασίζεται σε τρεις πυλώνες. Κωδικοποίηση και απλοποίηση των διοικητικών και νομικών διαδικασιών, επιτάχυση των σχετικών διαδικασιών, κάτι που εξυπηρετεί τόσο το στόχο της ε, συμμόρφωσης με τις δεσμεύσεις που έχει η Ελλάδα, όσο και το στόχο της καλύτερης προστασίας των ίδιων των ετούντων άσυλο και μέρημνα για τους πρόσφυγες που βρίσκονται στην Ελλάδα σύμφωνα τόσο με τις διεθνείς υποχρεώσεις της Ελλάδας όσο και τις αξίες μας. Βέβαια ο νόμος δεν λύνει από μόνος του όλα τα ζητήματα. Χρειάζονται μια σειρά διοικητικέ ενέργειες και πράξεις. Γι' αυτό το λόγο αυξάνουμε κατά 400 άτομα τους, ε, το προσωπικό της υπηρεσίας ασύλου και αυξάνουμε από 12 σε 20 ε, μέσα στο 2018 τις επιτροπές προσφυγών για να τις κάνουμε 30 το 2019. Ένα κύριο ζήτημα που αντιμετωπίσαμε αυτό το χρονικό διάστημα και ελπίζω οριστικά τα ήταν το ζήτημα της διερμηνία. Δεν θα μπω σε περισσότερε ε, ε, λεπτομέρειες. Αν ερωτηθώ θα σας πω περισσότερα. Τέλος, καταβάλουμε προσπάθειες για τη βελτίωση των συνθήκων υποδοχής ώστε να ανταποκριθούμε στι ε, ανάγκες που δημιουργούν οι ροέ. σε αυτό το πλαίσιο αναθεωρήσαμε και τον πρακτικό και τον οικονομικό προϋπολογισμό για το δεύτερο εξάμεινο του 2018 καταθέσαμε επικαιροποιημένο financial plan προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και καταθέτουμε στις επόμενες μέρες και νέο για το 2019. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα έχουμε ανθρώπους σε 27 εποπτευόμενες από την πολιτεία δομές και προχωράμε σε άνοιγμα 7 νέων δομών μέσα του προγράμματος Εστία φιλοξενούμε σε διαμερίσματα 21.000 άτομα μαζί με την ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ και θέλουμε να φτάσουμε τις 30.000 μέχρι το τέλος του 2018. Είχαμε 300 θέσεις για συνόδευτα ανήλικα. Αυτή τη στιγμή έχουμε 1.956 θέσεις και ο στόχος μας είναι να φτάσουμε τις 3.000 ε, θέσεις. Στόχος μας είναι μέσα τον Ιούλιο να μεταφερθούν στην ενδοχώρα 2.000 ευάλωτοι που, έχουν, που αυτή τη στιγμή βρίσκονται στα νησιά και συγχρόνως ε, τα νησιά τέλος του Σεπτεμβρίου να μην έχουν πάνω από 10.000 ανθρώπους. Οι ανήλικοι πρόσφυγες και μετανάστες εγγράφονται υποχρεωτικά στα δημόσια σχολεία, όπως και τα Ελληνόπουλα, σε ειδικές τάξεις υποδοχής, σύμφωνα με το σχεδιασμό που έχει το Υπουργείο Παιδείας. Τέλος, ξεκινήσαμε ένα πρόγραμμα ένταξης, το οποίο πάει πάρα πολύ καλά. Ολοκληρώνεται το πιλωτικό πρόγραμμα στη Λιβαδιά και στη Θήβα και στη Θεσσαλονίκη. Έχει τρία παραμέτρους, την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, τον προδιορισμό των δεξιοτήτων των προσφύγων και την πρόσφαση στην αγορά ε, εργασίας. Η πρότασή μας, η καινούργια μας πρόταση, είναι να δημιουργηθεί ένα ενδιάμεσο πρόγραμμα για αυτούς που πλέον έχουν πάρει άσυλο, με 5.000 ε, θέσεις για έξι μήνες και οι οποίοι θα εντάσσονται και στο ενταξιακό μας πρόγραμμα. Κυρίες και κύριοι, με μία έννοια αγαπητοί συνάδελφοι, η Ευρώπη βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι και αντιμέτωπη με μεγάλες προκλήσεις. Η αντίδρασή μας και η προσέγγισή μας στις προκλήσεις αυτές θα καθορίσουν το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις επόμενες γενιές. Ας θέλω να γίνω πιο σαφής. Δεν θα ορίσουν σε ποια πλευρά θα γυρίσει η Ευρώπη, αν θα γυρίσει προς την πλευρά των ανθρώπινων δικαιωμάτων και αξιών ή προς την πλευρά της, ε, αν θα γυρίσει προς την πλευρά δηλαδή της αλληλεγγύης ή προς την πλευρά της ξενοφοβίας και του ρατσισμού, δεν θα ορίσουν μόνο αυτό θα ορίσουν το μέλλον της Ευρώπης ως Ένωση. Θα πρέπει πάση θυσία να διαφυλέξουμε τις κοινέ μας ευρωπαϊκές αξίες, το σεβασμό στις κοινέ μας αποφάσεις, στις θυμελιώδες αξίες και στο διεθνές δίκαιο, στις αρχές της αλληλεγγύης και του ανθρωπισμού, στις οποίες βασίζεται το ευρωπαϊκό μας οικοδόμημα. Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ στα ειδικότερα αυτά θέματα, αλλά το τόσο σημαντικά για την πορεία της Ευρώπης και του κόσμου θέματα, είναι κέριος και σημαντικότερος από ποτέ. Γι' αυτό και ο ρόλος ο δικός σας, της κάθε μιας και του καθενός ξεχωριστά, είναι σημαντικός. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Υπουργέ. Τώρα θα ακούσουμε ερωτήσεις από τους βουλευτές. Να ξεκινήσω εγώ να σας ρωτήσω αναφέρατε ε, βεβαίως στη συνεργασία με τα κράτη της ε, πρώτης γραμμής να σας ρωτήσω αν ακούτε τίποτα για τις ε, προτάσεις του Δουβλίνου που δεν ευθυγραμμίζονται με αυτά τα οποία έχουμε πει ως θέση του Κοινοβουλίου που λέτε ότι και η Ελλάδα είναι κοντά σε αυτές. Παραδείγματος ε, κάποια κράτηση και η επεξεργασία ε, εκτός ε, ένωσης. Δεν ξέρω αν ακούτε κάτι ως μέλος του Συμβουλίου. Δεύτερον, ως διαχειριστική αρχή του προϋπολογισμού, πού βρισκόμαστε ως προς αυτό. Ξέρω ότι θα ακολουθήσουν και πιο λεπτομερείς ερωτήσεις. Λοιπόν, ξεκινάμε με τον κατάλογο. Και παρακαλώ δύο λεπτά ο καθένας. Κύριε Λόπης Αγγιλάρ. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ που ήρθατε, ευχαριστώ που μιλήσατε και σας ευχαριστώ για την ελληνική προσπάθεια να αντιμετωπιστεί αυτή η συνεχιζόμενη κατάσταση. Δεν είναι η ώρα για λόγους και ομιλίες. Έχουμε πολλά τέτοια ακούσει στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά τη διάρκεια της ε, μεταναστευτικής κρίσης. Τώρα είναι η στιγμή να δούμε κάποιες, ε, κάποια συγκεκριμένα θέματα, να απευθύνουμε συγκεκριμένες ερωτήσεις σε έναν υπουργό που έχει μια έδρα στο Συμβούλιο, που βρίσκεται το πρόβλημα. Γιατί σωστά το είπατε, εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπάρχει μια συμμαχία για να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση και να υπάρξει κάποια αλλαγή. Γιατί η αντίδραση μέχρι τώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και εννοούμε το Συμβούλιο είναι αποτυχία. Το ερώτημα είναι πώς ε, βλέπετε την πιθανότητα πριν το τέλος αυτής της ε, θητείας να υπάρξει κάποια συμμαχία εντός του Συμβουλίου για να ξεμπλοκαριστεί ε, όλη αυτή η κατάσταση από το τωρινό status quo του συστήματος ασύλου, δηλαδή το Δουμπλίνο, η κοινή ευθύνη. Ποιε είναι οι πιθανότητες της Ελλάδα, μαζί με κάποια κράτη-μέλη, με τη νέα κυβέρνηση της Ισπανίας, να προωθήσουν αυτό το οποίο αναμένουμε, γιατί τώρα έχει μπλοκάρει ο κανονισμός του Δουβλίνου και αυτό σημαίνει ότι όλο το σύστημα ασύλου έχει μπλοκάρει ότι δεν υπάρχει πρόοδος ούτε στις διαδικασίες υποδοχής, ε, στην εγκατάσταση, σε οποιοδήποτε νομοθέτημα αναμένουμε από το σύστημα ασύλου. Δεν γίνεται κανένα βήμα γιατί έχει μπλοκάρει ο κανονισμός του Δουβλίνου. Υπάρχει λοιπόν πιθανότητα πριν το τέλος της ε, θητείας να γίνει κάποια αλλαγή. Και τι βοήθεια μπορεί να σας δώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να υπάρξει αλλαγή στο Συμβούλιο. Λοιπόν, θα ακούσουμε τους συναδέλφους με τη σειρά που ζήτησαν το λόγο. Μπάρμπαρα Σπινέλη. Δύο λεπτά παρακαλώ. Ε, να ευχαριστήσω και εγώ πολύ τον Υπουργό Βίτσα και την Ελλάδα για τις προσπάθειες που κάνει εδώ και χρόνια σε πάρα πολύ δύσκολες ε, οικονομικές συνθήκες. Αυτό το οποίο θα ήθελα να ρωτήσω αφορά το σχέδιο κειμένου που έχουμε για μια πιθανή συμφωνία του Συμβουλίου για το Δουβλίνο γίνεται σαφής αναφορά σε μια ε, πολιτική εξωτερήκευση της πολιτικής ασύλου και πιο συγκεκριμένα για πλατφόρμες ε, ε, περιφερειακές στις οποίες αποβιβάζονται οι πρόσφυγες σε συνεργασία με την Υπατιαρμοστία για τους πρόσφυγες. Ουσιαστικά πρόκειται για κέντρα, για hot spots εκτός Ευρώπης. Θα ήθελα να γνωρίζω τη θέση της Ελλάδος επ' αυτού. Εγώ διαβλέπω μεγάλο κίνδυνο σε μια τέτοια πολιτική, διότι οι διαδικασίες ε, ε, μέσω των οποίων γίνεται διάκριση των προσφύγων με τους οικονομικούς ε, μετανάστες δεν είναι σαφής, δεν ξέρουμε με ποια κριτήρια θα γίνονται, δεν ξέρουμε αν αυτές οι τρίτες χώρες έχουν κατάλληλη νομοθεσία και αν θα δεχτούν ε, τις πλατφόρμες, ε, δεν αναφέρεται πολιτική επανεγκατάσταση resettlement, δεν αναφέρεται σε χώρες οι οποίες είναι λίγο πολύ ασφαλείς όσον αφορά το το διεθνές δίκαιο. Επομένως θα ήθελα να ξέρω ποια είναι η θέση της Ελλάδος, τι στάση θα τηρήσει και ε, σε τι συμμαχίες θα στοιχηματίσετε Δεδομένου ότι κατά πάσα πιθανότητα θα υπάρχει υποστήριξη της Ισπανίας, αλλά δεν θα υπάρχει στήριξη ε, από την Ιταλία που είναι και αυτή η χώρα πρώτης ε, άφηξης. Ε, δυστυχώς δεν θα έχετε τη στήριξη της Ιταλίας να προσθέσω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Μπάρμπαρα. Η κυρία Παγκαθαραουρτουντούα. Η κυρία Παγκαθαραουρτουντούα. Ζητώ συγγνώμη. Επειδή το επίθετό μου είναι τόσο δύσκολο, ξέρετε ότι δύσκολα μπορώ να καταλάβω ότι απευθύνεστε σε μένα. Το μαθαίνω λίγο καλύτερα, λέει ο πρόεδρο. Σιγά σιγά. Βελτιώνεστε, βελτιώνεστε, αλλά ήμουν λίγο αφιερωμένη. Ζητώ συγγνώμη. Καταρχά, ε, να ευχαριστήσω πάρα πολύ για την ε, παρουσία σα εδώ και σας ε, ευχαριστώ διότι πράγματι εσείς έχετε δίκιο. Πρέπει να καθορίσουμε το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχετε δίκιο σε όσα είπατε η Ελλάδα έχει αναλάβει ένα από τα πιο σημαντικά καθήκοντα και ε, εμείς αν έχουμε κοινά σύνορα, έχουμε κοινά σύνορα και αν πρέπει να υπάρχουν κοινέ προκλήσεις πρέπει να αντιμετωπίσουμε από κοινού. Δεν μπορούμε να αφήσουμε εσά ε, με όλο το βάρος ε, της ε, αντιμετώπισης κατάστασης. Ε, πρέπει όμως να προβάλλουμε και τα στοιχεία σε κάθε χώρα μας. Αναφέρατε τους αριθμούς, διότι πολλά πράγματα είναι κρυφά. Η κοινή γνώμη ε, δεν ασχολείται όπως ασχολιόταν το 2015 ή το 2016. Επομένως, θα ήθελα να σας ρωτήσω τι εθνικότητες ε, έχετε κατά προτεραιότητα στην Ελλάδα τι ποσοστό ανηλίκων, πέραν των όσων μας είπατε ότι θέλετε να φτάσετε ε, σε σχέδια υποδοχής 3.000 ε, ε, ασυνόδευτων ανηλίκων. Πόσοι είναι. Επίσης αναφερθήκατε στα σχολεία και είπατε ότι αυτά τα ανήλικα παιδιά μπορούν να πάνε στο σχολείο, αλλά πόσα πηγαίνουν στο σχολείο αυτή τη στιγμή, σε τι ποσοστό. Και επίσης αναφερθήκατε και στην ανάγκη να ε, ξεκινήσουν αυτή οι τριμερής διάλογοι με το Συμβούλιο και εμείς είμαστε μαζί σας. Δώστε μας όμως τα απαραίτητα ε, μέσα για να μπορέσουμε και εμείς να προβάλλουμε την κατάσταση και να μην αφήσουμε ε, την Ελλάδα να αντιμετωπίσει μόνη της την κατάσταση. Κατά τα λοιπά, αναφερθήκατε στην κατάσταση στα νησιά και τα προβλήματα που αντιμετωπίζονται. Ε, πώς μπορούμε λοιπόν να σας βοηθήσουμε και σε αυτό δώστε μας κάποιες ενδείξεις, διότι εμείς δεν παίρνουμε όλες τις πληροφορίες. Εκμεταλλευτείτε λοιπόν αυτή την ευκαιρία και δώστε μας και την όθηση που χρειαζόμαστε για να μπορέσουμε και εμείς να σας βοηθήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κύρκος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, καταλαβαίνετε πως η παρουσία σας εδώ σήμερα είναι πολύ σημαντική. Κυρίως για αυτά που είπε και η τελευταία συνάδελφος. Ε, μας λείπουν πληροφορίες. Στην Επιτροπή, ξέρετε, από όλε τι πλευρέ ε, βρίσκεται συμμάχο. Αλλά χρειαζόμαστε πληροφορίε σε περισσότερο βάθο από αυτά που μα δίνει η Κομισιόν. Γιατί μόνο έτσι μπορούμε να προχωρήσουμε και εμεί σε στήριξη και συγκεκριμένων δράσεων και να ενημερώσουμε και το κοινό μα, τι χώρε μα, για το τι ακριβώ γίνεται στην Ελλάδα. Μία μικρή ερώτηση. Μέρκελ Μακρόν. Χθε μα μιλήσανε πολύ για να σταματήσουν τα ρεύματα των παράνομων μεταναστών. Δεν είπαν τίποτα για τους πρόσφυγες, δεν είπαν τίποτα για το κοινό σύστημα ευρωπαϊκού ασύλου. Τι πιστεύετε ότι θα γίνει με αυτό. Και δεύτερο, αν δεν γίνει με τη Βουλγαρική Προεδρία, τι ελπίδες έχει να γίνει με την Αυστριακή οτιδήποτε για το Δουβλίνο και το πακέτο των πραγμάτων. Ευχαριστώ. Okay, Ο Μίλτος έθεσε την ερώτηση, αλλά ήταν πιο σαφής ε, την ίδια ερώτηση ε, ε, που έθεσα κι εγώ. Η κυρία Κέγκε στη συνέχεια. Ευχαριστώ και εγώ ε, τον Υπουργό, ε, τον κύριο Βίτσα, για την παρουσίασή του. Συμφωνώ πολύ ε, με την ανάλυση σας για τις κοινέ αξίες και την εκτίμηση των κοινών στόχων που πρέπει να επιτύχουμε. Η δημιουργία ενός κοινού συστήματος ασύλου, το οποίο θα έχει αλληλεγγύη και θα σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εμείς από πλευράς Κοινοβουλίου θα κάνουμε ό,τι μπορούμε και θα πιέσουμε. Στην πραγματικότητα πιέζουμε ήδη και έχουμε ξεκινήσει από όλε τις προτάσεις που παρουσιάσατε που περιλαμβάνονται στην ολιστική προσέγγιση που ψήφισε με πολύ μεγάλη πλειοψηφία τον Απρίλιο του 2016 το 2016 και μετά τον Νοέμβριο του 2017 υπερασπιζόμαστε τη θέση που εγκρίναμε που είναι η μόνη η οποία προτείνει ένα ισότιμο σύστημα ασύλου. Πρέπει να βρούμε ένα κοινό σύστημα αλλά επί βάσεως. Έχετε δίκιο σε αυτό αλλά επί βάσεως. Η πρόταση της Βουλγαρικής Προεδρίας γιατί αυτήν συζητούμε ή τη βάση των ε, τελευταίων δηλώσεων που διαβάζουμε διαβάσαμε στον τύπο για προτάσεις οι οποίες κατά την άποψή μου είναι τοπικές. Προβλέπουν ε, περιφερειακές πλατφόρμες για να γίνεται διάκριση μεταξύ οικονομικών μεταναστών και αυτών που κάνουν αίτηση ασύλου για διεθνή προστασία για να μην ε, μπορέσουν να φτάσουν εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, εγώ πιστεύω ότι εσείς που βρίσκεστε στο Συμβούλιο θα πρέπει να πάτε εκεί και να μιλήσετε με τα κράτη-μέλη να παρουσιάσετε τις ε, θέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, από τη μια την πρόταση του Δουβλίνου η οποία ψηφίστηκε με πολύ μεγάλη πλειοψηφία τον Οκτώβριο του 2017 και από την άλλη όλα τα σημεία τα οποία αφορούν την ολιστική προσέγγιση. Να μην έχουμε απλώς ένα σημείο, αλλά όλα τα σημεία στα οποία αναφερθήκατε. Νόμιμες οδοί, ε, πώς μπορούμε να κάνουμε παρέμβαση στα βαθιά, ε, βαθύτερα αίτια. Εγώ πιστεύω ότι δεν λείπουν προτάσεις, λείπει η πολιτική βούληση και αυτό ζητούμε. Και αυτό είναι και το μήνυμα το οποίο θα πρέπει να δοθεί στην επόμενη Προεδρία. Yes, colleagues have been asking what is the scope for you getting Πολλοί από τους ε, συναδέλφους φαίνεται ότι ρωτούν για το τι πρόκειται να συμβεί στο Συμβούλιο. Φαίνεται ότι ανησυχούν. Κύριε Βόνμπεργκ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ. λέγεται ότι έχει μειωθεί ο αριθμός των μεταναστών που έρχονται στην Ελλάδα, το αριθμός των αφήξεων. Όμως, έχει υπάρξει συνολικά από χρόνο σε χρόνο αύξηση. Και αυτό που δεν καταλαβαίνω εγώ είναι γιατί συμβαίνει αυτό δεδομένου ότι είχαμε τη συμφωνία με την Τουρκία. Υποτίθεται ότι η συμφωνία με την Τουρκία θα είχε μειώσει ε, αυτές τις ροές και ότι υπήρχε μια συμφωνία μάλιστα για επιστροφές ένας προς έναν. Πόσοι ε, απεστράφησαν στην Τουρκία επί τη βάση της συμφωνίας θα ήθελα εγώ να ρωτήσω. Είδαμε πρόσφατα στον τύπο ότι συνέβη με το πλοιάριο του Κουάριους που προσπαθούσε να βρει λιμάνι που πέρασε από την Ιταλία που δεν το δέχτηκε η Μάλτα και κατέληξε στην Ισπανία παρόλο που γνωρίζουμε ότι και η Ισπανία δεν έχει τις ε, υποδομές και τη δυνατότητα να υποστηρίξει αυτούς τους νεοφυχθέντες. Μήπως θεωρείτε ότι μετά από αυτές τις εξελίξεις θα αποφασίσουν περισσότεροι να στραφούν προς τα ελληνικά νησιά. Δηλαδή, αν η μία χώρα μετά την άλλη στην Ευρώπη αρχίζουν να αρχίζει να αρνείται να εφαρμόζεται ένα σύστημα ασύλου που προσπαθήσαμε να χτίσουμε επί χρόνια, ε, το ερώτημα που έχω εγώ είναι πόσα χρόνια ακόμα, πόσον καιρό ακόμα θα μπορέσει η Ελλάδα και ο πληθυσμός της να αντιμετωπίζει όλους αυτούς τους μετανάστες που έρχονται στη χώρα. Της, στη χώρα έχω ακούσει, έχουμε ενημερωθεί από τον τύπο ότι έχουν υπάρξει και επεισόδια και συγκρούσεις ανάμεσα σε μετανάστες που βρίσκονται στα κέντρα υποδοχής και στον τυπικό πληθυσμό. Ε, ή επίσης και στην ενδοχώρα μπορεί κάποια στιγμή να έχουμε αντίστοιχα ε, επεισόδια. Επίσης η επόμενη προεδρία του Συμβουλίου είναι η Αυστρία και από όσο γνωρίζω έχει κάποιες πολύ διαφορετικές προτάσεις ε, σε σχέση με το πώ θέλει να αντιμετωπίσει την μετανάστευση τη μετανάστευση γενικότερα. Σα ευχαριστώ. Και αφού σα καλωσορίσω και εγώ με τη σειρά μου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ε, θα ήθελα να σας ρωτήσω για τη θέση σας σε σχέση με τα όσα ακούγονται ε, τις τελευταίες ημέρες από τη Γερμανία, όπου, όπως θα γνωρίζετε, απειλείται η ίδια η κυβερνητική σταθερότητα λόγω της ε, πρόθεσης, όπως λέγεται τουλάχιστον, του Γερμανικού Υπουργείου Εσωτερικών να αξιώσει επαναπροωθήσεις ετούντων άσυλο προς τις χώρες πρώτης υποδοχής προκειμένου να μειωθεί ο φόρτος τον οποίο, ο οποίος υπάρχει κατά τη γνώμη του Γερμανού Υπουργού Εσωτερικών στην Γερμανία. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω εάν τυχόν μπορούσαν να υλοποιηθούν τέτοιες προθέσεις, ειδικότερα σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, για επαναπροωθήσεις από τη Γερμανία προς την Ελλάδα, ποιες θα ήταν οι συνέπειες για την Ελλάδα και μήπως αυτό θα δημιουργούσε συνθήκες ανθρωπιστικής κρίσης με απρόβλεπτες περαιτέρω συνέπειες, τις οποίες ενδεχομένως δεν θα μπορούσε και να τις αντιμετωπίσει με τα δικά του πενιχρά μέσα το ελληνικό κράτος. Ευχαριστώ. Thank you, Ellie. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, σα ευχαριστώ που εκφράσατε την υποστήριξη τη ελληνική κυβέρνηση, στη φιλόδοξη μεταρρύθμιση του κανονισμού του Δουβλίνου που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά από μια πολύ λεπτή και σημαντική διαπραγμάτευση. Η μεταρρύθμιση είναι πάρα πολύ σημαντική και δημιουργεί το μοναδικό ευρωπαϊκό σύστημα στο οποίο υπάρχει επιμερισμό των ευθυνών και ακυρώνει ε, την άδικη ε, διαδικασία τη χώρα ε, υποδοχή υποδοχή και ξεκινά μια διαδικασία που βάζει βάζει στο επίκεντρο του ανθρώπου, καθορίζει του σημαντικού του δεσμού και εξασφαλίζει ότι κάθε ευρωπαϊκή χώρα συμμετέχει στην υποδοχή. Ανησυχούμε, κύριε Υπουργέ, που στι 28 του μηνό ε, το Συμβούλιο θα αποφασίσει για άλλη μια φορά να μην αποφασίσει τίποτα. Είναι ε, αδιανόητο να μην έχει βρεθεί καμία λύση για την εσωτερική αλληλεγγύη και να μην έχουν λάβει καθόλου υπόψη τι προτάσει που υπερψήφισε τα δύο τρίτα του Κοινοβουλίου. Έχετε μια ιστορική ευθύνη στι 28 Ιουνίου να αποφασίσετε για το Διβουλίνο. Και αν οι κυβερνήσεις χάσουν αυτή την ευκαιρία, δεν θα πρέπει να έχετε ψευδεστήσει ότι θα διασώσετε το ευρωπαϊκό όραμα. Η αδράνεια και η ανικανότητα ε, να δοθούν απαντήσει σε προκλήσει οι οποίε είναι σαφώ κοινέ, ε, είναι αυτέ οι οποίε έχουν ανοίξει ε, τις πόρτε των φασιστικών και των λαϊκιστικών προκλήσεων στι χώρε μα. Πρέπει λοιπόν να δώσετε το βήμα για την αλληλεγγύη στην οποία εδράζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν πιστεύετε ότι θα κλείσετε μια ολόκληρη θάλασσα, πραγματικά απατάστε ικτρά. Πρέπει να υπάρχουν πολιτικέ εξωτερήκευση ε, των ε, συνόρων μα. Μην θεωρείτε ότι είναι πρώτη πρωτότυπο, δεν είναι τίποτα καινούριο. Το δοκίμασαν όλοι εδώ και χρόνια, ποτέ δεν λειτουργήσε ένα τέτοιο σύστημα και πάντα ανοίγουν νέε διαδρομέ, οι οποίε είναι πιο ε, επικίνδυνε ακόμα προ την Ιταλία και προ την Ελλάδα. Χρειάζεται ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και νόμιμε οδοί πρόσβαση σε όλε τι ευρωπαϊκέ χώρε. Στι 28 το Συμβούλιο πρέπει να συζητήσει και να αποφασίσει και σας ζητώ να κάνετε ό,τι μπορείτε, ό,τι περνάει από το χέρι σα, προκειμένου στι 28 να μην χαθεί αυτή η ιστορική ευκαιρία, διότι γι' αυτό το θέμα είμαι πεπισμένη ότι διακυβεύεται το ίδιο το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ πολύ. Thank ε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Τζέζεκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ ένα think tank η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Σταθερότητας με έδρα το Βερολίνο και ο πρόεδρος του είναι ο Γκέρχαρτ Νάους. Θα θυμάστε ότι ήταν οι αρχιτέκτονες της ιδέας της συμφωνίας μεταξύ Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για να διαχειριστούμε τις μεταναστευτικές οδούς που οδηγούν ε, και στην Ελλάδα τώρα προτείνουν μία άλλη ιδέα για το πώς θα αντιμετωπίσουμε την διαδρομή απόλυτη και το βασικό στοιχείο είναι να επιταχυνθεί η διαδικασία ασύλου όπως στην Ολλανδία που χρειάζονται δύο μήνες για την επεξεργασία και προσφυγή και τα λοιπά όλα και θεωρούν ότι αν ισχύσει αυτό στις νότιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μαζί με συμφωνίες επιστροφής τότε βεβαίως ε, θα υπάρξει διάκριση μεταξύ αυτών που όντως ε, ετούνται άσυλο και λοιπόν ε, θα ήθελα να μάθω λοιπόν την άποψή σας για αυτήν την ιδέα και τι βοήθεια ή μέτρα θα απαιτούσε από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να προσπαθήσετε να το επιτύχετε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Μαρτίνα Άντερσεν. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ για τις ε, πληροφορίες ε, και νομίζω πως ε, πολλοί από μας εδώ πέρα θα συμφωνήσουμε ότι κανείς δεν θέλει να γίνει πρόσφυγας και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, να ευχαριστήσω την Ελλάδα για τις προσπάθειες που κάνει παρά το ότι δεν υπάρχουν ε, ασφαλείς ε, και νόμιμες ε, διόδοι και δεδομένες της ημέρας είναι ενδιαφέρον ότι έχουμε και μία συνάντηση κορεπέρ και προκύπτουν διάφορες πληροφορίες για τα hot και την εξωτερική ανάθεση των συνόρων που είναι σοκαριστικό και καμιά φορά ξεχνάμε εδώ μέσα την λέξη αλληλεγγύη. Ε, υπάρχει μόνο η αλληλεγγύη των αποθήσεων και φαίνεται ότι έχει γίνει αποδεκτό. Σιγά σιγά έρχεται στο τι θα πρέπει να γίνει. Και υπάρχει αυτή η μάχη των αξιών που αναφέρατε, που χάνεται το διεθνές δίκαιο που έχουμε στην Γενέβη, το πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης, όλα αυτά αγνοούνται. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω, κυρίως για το θέμα της διακίνησης και των διακινητών στην Ελλάδα και αλλού ε, στην Ευρώπη. Τι πρόοδο και τι προκλήσεις έχετε κάνει όσον αφορά και την ε, ένταξη. Είπατε από τον Απρίλιο πάνω από 6.500 άτομα έχουν έρθει στην Ελλάδα είτε πρόσφυγες είτε οικονομικοί μετανάστες από τη φτώχεια και την κλιματική αλλαγή και το θέμα βεβαίως της οικογενειακής επανένωσης να αναγνωρίσουμε και τα πρακτικά και νομικά εμπόδια που υπάρχουν. Και θα ήθελα και πάλι να σας ευχαριστήσω για όλες τις ε, προσπάθειές σας και πρέπει να σας στηρίξουμε να κάνετε περισσότερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η κυρία Βόζενμπεργκ. Κύριε Υπουργέ, ευχαριστούμε που ήρθατε στην Επιτροπή μας να μας ενημερώσετε. Ε, υπόθηκε πριν από συνάδελφο το ένα καινούριο δεδομένο ότι η κυρία Μέρκελ, η Γερμανία, πιέζεται από το Υπουργείο Εσωτερικών, από τον κύριο Ζέχοφερ, να ε, ε, ε ενεργοποιήσει την πρόβλεψη του Δουβλίνου για επιστροφές στις πρώτες χώρες υποδοχής ε, προσφύγων. Παράλληλα όμως ξέρουμε ότι η Γερμανία έχει παγώσει τη διαδικασία των οικογενειακών επανενώσεων με αποτέλεσμα να υπάρχουν μέλη οικογενειών τα οποία είναι διάσπαρτα στα κράτη-μέλη και ιδιαίτερα στη χώρα μας πολλά ως, ε, με το δεδομένο ότι είναι χώρα πρώτης ε, εισόδου. Θέλω να σας ρωτήσω κατά πόσον η κυβέρνηση της Ελλάδος αυτό το θέμα το έχει αναδείξει ή πώς πρόκειται να το διαχωριστεί δεδομένου ότι και αυτό είναι μια πρόνοια που υπάρχει στο ισχύ Αρχείων μέχρι σήμερα Δουβλίνο. Σας ευχαριστώ πολύ. Στον κανονισμό εννοώντας. Thank you. And please. παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, δεν θα επαναλάβω και πάλι το ότι η μεγάλη πλειοψηφία των ε, μεταναστών και προσφύγων φιλοξενείται σε τρίτες χώρες εκτός της Ένωσης, αλλά θα επιμένω πάντα για να είναι και η Ευρωπαϊκή Ένωση ένας χώρος υποδοχής και ένταξης ανθρώπων που φεύγουν από πολιτικές διώξεις και βασανιστήρια. Και είναι κρίμα αυτό το οποίο βλέπουμε τώρα στη Γερμανία, γιατί το να τους ε, στέλνουμε όλους πίσω χωρίς να μιλάμε για μετεγκατάσταση σημαίνει ότι όλη η πίεση πέφτει σε κάποιες χώρες με εξωτερικά σύνορα. Είναι ευρωπαϊκή λύση. Ε, το είπατε σαφώς. Η ευρωπαϊκή λύση υπάρχει. Βρίσκεται εδώ, βρίσκεται στο Κοινοβούλιο, αναφέρατε κάποια σημεία που αφορούν την μετεγκατάσταση, νόμιμους τρόπους ε, όπως η μετεγκατάσταση και η μπλε κάρτα και μια νέα συνεργασία με τις χώρες προέλευσης για να διασφαλίσουμε ότι ε, λιγότεροι άνθρωποι θα παρασύρονται από ψεύτικες υποσχέσεις ε, των λαθροδιακινητών ε, και οι χώρες θα είναι σε θέση να υποδεχτούν ξανά και να επανεντάξουν τους πολίτες τους. Παρ' όλα αυτά τώρα βρισκόμαστε στην ε, σημερινή μα κατάσταση και η τένεια που και η εισαγωγή σα δείχνουν ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει μεγάλε προκλήσει, αλλά η κατάσταση εξελίσσεται και εργάζεστε σε μια περίπλοκη κατάσταση. Όσον αφορά την κατάσταση στα νησιά, θα ήθελα να κάνω κάποιες συγκεκριμένες ερωτήσεις. Αναφέρατε τα 60.000, τα 16.000 άτομα στα νησιά και είπατε ότι προσπαθείτε να μειώσετε αυτούς τους αριθμούς. Μπορείτε να μας εξηγήσετε τι σημαίνει αυτό. Θα στείλετε περισσότερους ανθρώπους στην Τουρκία ή με την κατάσταση βελτιώνεται. Μήπως θα βάλετε περισσότερους ανθρώπους ε, στην ε, υπηρετική χώρα. Και τι γίνεται με την στήριξη που λαμβάνετε από την ε, Κομισιόν ε, ή άλλα κρατημέλη για την ένταξη. Μπορείτε να μας πείτε κάποια περισσότερα πράγματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μπίργκιτ. Δεν θέλει κάποιος άλλος να μιλήσει. Ωραία. Λοιπόν, θα σας το πω τώρα γιατί δεν θα ακουστεί όταν ε, τελειώσετε. Ε, πολλοί συνάδελφοι εδώ εργάζονται πάνω σε αυτά τα θέματα Δουβλίνου βεβαίως. Ε, γι' αυτό ακριβώς ε, ε, και εσείς ως μέλος του Συμβουλίου, γιατί αυτά εξαρτώνται από το Συμβουλίο, από το Συμβουλίο δέχεστε τόσες πολλές ερωτήσεις ειδικά σήμερα, την μέρα των προσφύγων. Οπότε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο, έχετε και αρκετό χρόνο για να απαντήσετε στις ερωτήσεις. Ε, ευχαριστώ για τις ερωτήσεις που δείχνουν από διάφορες οπτικές ε, γωνίες την, ε, το ενδιαφέρον. Το ενδιαφέρον για την εξέλιξη του προσφυγικού μεταναστευτικού ζητήματος. Ε, θα ήθελα όμως να επισημάνω πριν απαντήσω μία-μία τις ερωτήσεις ορισμένα ε, στοιχεία που τα έχουμε υπόψη μας. Γνωρίζουμε πόσοι πρόσφυγες αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην Ιορδανία. Έξι εκατομμύρια. Έξι εκατομμύρια. Πόσοι πρόσφυγες βρίσκονται στην Τουρκία. Τρία εκατομμύρια. Ε, καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν χώρες που διαχειρίζονται, αυτό θέλω να πω, πολύ μεγάλα ε, προβλήματα. Και πριν απαντήσω σε ερωτήσεις, θέλω να σας πω ότι μου γεννήσατε μια πάρα πολύ καλή ιδέα που μου την είπαν και Έλληνες ευρωβουλευτές εχθές ε, και νομίζω ότι πρέπει να την ξεκινήσουμε, ε, δικιά μας ευθύνη είναι σαν ελληνική κυβέρνηση, να υπάρχει ένα μηνιαίο ήδη μηνιαίο report ε, προς τους ευρωβουλευτές της ΛΥΜΠΕ μέσω είτε απευθείας από το Υπουργείο είτε μέσω της μόνιμης αντιπροσωπείας της Ελλάδας ε, στην, ε, Βρυξέλλες ώστε πραγματικά να έχετε την, τουλάχιστον τη δική μας πλευρά ε, ενημέρωσης. Γιατί πολλές φορές όλοι μας βρισκόμαστε, και θα <laughs> αναφερθώ και σε αυτό, ε, μπροστά στο ότι έχουμε την πληροφόρηση μόνο από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δεν θέλω να τα κρίνω, αλλά μερικές φορές άλλο είναι το ένα, άλλο είναι το άλλο. Και μακάρι να μπορέσουμε να κάνουμε και άλλου είδου ε, συνεργασίες ώστε να έρθουν εδώ και άνθρωποι του πεδίου. Τι εννοώ άνθρωποι του πεδίου. Εγώ είμαι υπουργό. Γύρω μου είναι συνεργάτες σε ένα επίπεδο. Υπάρχουν άνθρωποι όμως που καθημερινά δουλεύουν με τους πρόσφυγες. Δουλεύουν στα ΚΑΜΠ, κάνουν καταγραφές, κάνουν διερμηνίες. Και εγώ προσπαθώ να μάθω πολλοί από αυτούς πηγαίνοντας εκεί. Και όχι από τη σιγουριά, αν θέλετε, του γραφείου. Γιατί εκεί στη μάχη φαίνονται και τα προβλήματα. Τώρα, να πω μερικά γρήγορα για την Ελλάδα. Αυτό θα σας στείλω και όλο το πληροφοριακό ε, υλικό σε σχέση με τις ερωτήσεις και να καπιαστώ λίγο περισσότερο με το, τις εξελισσόμενες διαδικασίες για το Δουβλίνο 4 και άλλες ιδέες, θα έλεγα εγώ. Δουβλίνο 4 και άλλες ιδέες που ακούγονται γύρω-γύρω η Ελλάδα έχει απορροφήσει σε σχέση με το εθνικό της μέλος το 30% μέχρι το τέλος του 2017 των παρεχόμενων χρημάτων από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Κομισιόν. Το, ποσοστό, το, το, πρόγραμμα είναι μέχρι το 2020. Δεν έχουμε εγγραφές του, 2000, του τέλους του 2017 ε, και δεν έχουμε και εγγραφές του 2018 για να σας δώσω περισσότερα στοιχεία. Δύο πράγματα θα σας πω. Το ένα ότι ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση απορρόφησης είναι 10%. Αλλά δεύτερο πράγμα πρέπει να σας πω, προσπαθούμε να τα καταφέρουμε καλύτερα. Δηλαδή θεωρούμε ότι οι διαδικασίες που έχουμε είναι αρκετά αργές και μας λείπουν χρήματα με την έννοια ότι υπάρχουν τα χρήματα και δεν τα έχουμε ακόμα χρησιμοποιήσει στο πεδίο για τους πρόσφυγες. Αυτό τώρα θέλει μια σειρά αλλαγές. Το 2015 δεν είχαμε Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Υπήρξε, δεν είχαμε διαχειριστική αρχή αυτών των ε, χρημάτων. Θέλω να σας πω ότι αυτά τα προβλήματα προσπαθούμε να τα λύσουμε και η κριτική μερικές φορές κάνει η πάντα για μένα, ακόμα και η κακοπροαίρετη κριτική, έχει τα καλά της στοιχεία. Δηλαδή, εγώ τη δέχομαι ώστε να προσπαθήσουμε ακόμα περισσότερο, ακόμα πιο έντονα. Η κούραση δεν είναι από τις οψιών που πρέπει να παίρνεις υπόψη σου και αυτό είναι το βασικό μας ε, ζήτημα. Περίπου εκεί είμαστε. Τι κάναμε τώρα. Είχαμε ένα προϋπολογισμό εγκεκριμένο το 2018 θεωρήσαμε στο τέλος του Μαρτίου ότι οι εκτιμήσεις μας που έγιναν το 2017 για το 2018 είχαν υποτιμήσει το τι θα συμβεί. Και στείλαμε στην Κομισιόν ένα αναθεωρημένο πρόγραμμα. Σας δίνω μία μόνο πλευρά. Με βάση την τότε ε, εκτίμηση θα έπρεπε στο τέλος του Ιουνίου να κλείσουμε 11 επιπλέον κέντρα φιλοξενίας η απόφαση μας ήταν να ανοίξουμε, να διατηρήσουμε αυτά τα 11 και να ανοίξουμε, έχουμε ανοίξει ήδη άλλα τρία και θα ανοίξουμε άλλα τέσσερα. Σας δίνω αυτό το παράδειγμα για να καταλάβετε τη ε, διαφορά. Αυτό, αυτός ο αναθεωρημένος προϋπολογισμός, έχουμε όλη την πληροφόρηση ότι μέχρι το τέλος του μήνα θα έχει εγκριθεί. Συγχρόνως προετοιμάζουμε ώστε να ολοκληρωθεί το Σεπτέμβριο ως απόφαση, εμείς το έχουμε ήδη έτοιμο, τον προϋπολογισμό του 2019. Τι θα συμβεί ανάμεσα στο 2018 και στο 2019, δεν θα υπάρξει έκτακτη βοήθεια. Δηλαδή, το κομμάτι της έκτακτης βοήθειας τελειώνει. Θα υπάρξει τακτική βοήθεια. Άρα μπαίνουμε εκεί και ενισχύεται και ο προϋπολογισμός του Υπουργείου. Αυτό είναι, αυτά είναι τα δύο βασικά ζητήματα. Σε τι προετοιμαζόμαστε, η τακτική βοήθεια, η DigiHome, έχει πιο δύσκολες διαδικασίες σε σχέση με την DigiEco, που έδινε τα χρήματα απευθείας σε διεθνείς ε, οργανισμούς. Άρα από τώρα πρέπει να προετοιμαστούμε ώστε ως το τέλος του χρόνου να έχουν λυθεί αυτά τα ζητήματα. Το έχουμε δηλαδή στο μυαλό μας. Άρα πρέπει να ξεπεράσουμε γραφειοκρατίες, διαδικασίες και να λειτουργήσουμε με τη λογική ότι η δουλειά που κάνουμε έχουν, έχει να κάνει με τους ωφελούμενους και δεν έχει να κάνει με τις... Άρα θέλουμε διαδικασίες υπέρ των ωφελουμένων και όχι διαδικασίες υπέρ των διαδικασιών. Πάντοτε με διαφάνεια, πάντοτε ε, με έλεγχο κτλ. Υπήρξα ε, αναπληρωτής υπουργός ε, εθνικής Άμυνας με... και μία από τις αρμοδιότητές μου ήταν ο συντονισμός ε, όλων των Υπουργείων για τη μετανάστευση. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας έχει συμβάλει πάρα πολύ. Ε, ενισχύθηκε από την έκτακτη χρηματοδότηση με περίπου 100 εκατομμύρια. Έγινε ο έλεγχος των 100 εκατομμύριων και πήραν το OK τα 99 εκατομμύρια 800.000. Δηλαδή η δουλειά έγινε και σωστά και ε, ωφέλιμα. Και αυτό, πρέπει να το ε, σπρώξουμε ε, παντού. Ε, το δεύτερο. Ε, δυστυχώς έχω λίγο χρόνο. μου ζητάνε να μιλάω πιο αργά, αλλά έχω λίγο χρόνο και κάνω... ναι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 ε, περίπου 40% είναι Σύριοι, περίπου 12 με 13% είναι Αφγανοί και Ιρακινοί, αυτά είναι τα, τα δύο δεύτερα μεγάλα ε, κομμάτια, και το τέταρτο κομμάτι είναι Πακιστανοί. Αυτές είναι, αυτά είναι οι, οι πολλοί. Αλλά θέλω να σας δώσω ένα... Στο, στο νέο budget έχουμε προβλέψει πάρα πολλά για τη διερμηνία. Είχαμε ένα μεγάλο πρόβλημα στις αρχές του 2018. Το λύσαμε αυτό το πρόβλημα. Αλλά θέλω να σας πω ότι χρειαζόμαστε διερμηνείς για 38 γλώσσες. Για να έχουμε μια αίσθηση. Δηλαδή στη Μόρια, στη Λέσβο, χρειαζόμαστε διερμηνείς για 38 γλώσσες. Να τα προβλήματα πια που μπαίνουν, που υπάρχουν στο πεδίο. Γενικά οι ανήλικοι στατιστικά είναι ανάμεσα στο 27 με 30% του συνολικού πληθυσμού. Εδώ πρέπει να κάνουμε μια διάκριση. Ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των, από τους ανήλικους είναι με τις οικογένειές τους. Ένα μικρότερο κομμάτι είναι ασυνόδευτοι οι ανήλικοι από αυτό το κομμάτι των ασυνόδευτων ανήλικων που είναι περίπου το 5% του συνολικού ε, πληθυσμού περίπου το 60 με 70% είναι ανάμεσα στα 15 και στα 18 χρόνια. Με βάση το νέο νόμο η φροντίδα των ανηλίκων περνάει στη Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής ε, Πρόνοιας. Και με αυτόν τον τρόπο χτίζουμε γρήγορα και μέσα ελπίζουμε μέχρι το τέλος του χρόνου να το έχουμε ολοκληρώσει 3.000 θέσεις φιλοξενίας με βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Σημασία για μας έχει κανένα παιδί, κανένας ανήλικος να μην βρίσκεται σε safe zone. Safe zone είναι ε, κομμάτια των ΚΑΜΠ όπου ξενούνται ξεχωριστά οι ασυνόδευτοι ανήλικοι, αλλά να είναι σε κανονικές δομές. Δεν θέλω να σκέφτομαι και κάθε φορά, τέλος πάντων γίνεται πάρα πολύ μεγάλος θόρυβος στο Υπουργείο, ότι μπορεί να υπάρξει ή κάθε φορά πρέπει να το κάνουμε πάρα πολύ γρήγορο γιατί όταν γίνεται, γίνεται για λόγους ασφαλείας, ανήλικο παιδί σε κρατητήριο. Αυτό πρέπει να ε, λυθεί και προηγούμενες καταστάσεις έχουν πια ε, ξεπεραστεί. Ε, πόσα τώρα πηγαίνουν στο σχολείο. Δεν είμαι, θα σας στείλω το, ε, δεν έχω αυτό το στοιχείο. Μπορώ όμως να σας πω ότι στον Ελαιώνα, ένα από τα μεγαλύτερα κάμπ στην Ελλάδα, αν δεν κάνω λάθος το δεύτερο μεγαλύτερο σε πληθυσμό, προχθές έγινε μια πολύ μεγάλη γιορτή των γύρω δημοτικών σχολείων, οκτώ δημοτικά σχολεία, τα οποία αυτά τα σχολεία είναι, ε, είναι και παιδιά ε, προσφύγων και μεταναστών και Ελληνόπουλα. Και πραγματικά ένιωθε κανένας άνθρωπος, πραγματικά η μετουσίωση της ανθρώπινης ουσίας πια, όταν ήταν σε αυτή τη γιορτή. Και πώς τη στήσανε οι δάσκαλοι και τα λοιπά. Ε, θα έχουμε κάποια ζητήματα γιατί με, υπάρχει ένας καταμερισμός σε σχέση με τα σχολεία και τώρα σε μερικά σχολεία θα πρέπει να γίνονται μεταφορές σε άλλες περιοχές γιατί δεν φτάνουν δηλαδή οι αίθουσε, αλλά είναι ζητήματα που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Ε, έχουμε συλλάβει 350 διακινητές την τελευταία χρονιά στην Ελλάδα. 350. Έλληνες, Ουκρανούς, ε, Τούρκους και πάει λέγοντας. Η μάχη ενάντια στους διακινητές πρέπει να είναι η πιο μεγάλη μάχη. Γνωρίζετε φαντάζομαι όλοι σας ότι από άποψη οικονομική, μετά την, ε, του, τους εξοπλισμούς, μετά τα ναρκωτικά, το τρίτο είναι η διακίνηση, η μετακίνηση ανθρώπων το τρίτο. Άρα είναι μια μεγάλη εγκληματική πράξη και η αστυνομία μας και σε συνεργασία και με άλλους πρέπει να βελτιωθεί, ε, όχι από την δική μας τη μεριά, από τον άλλον την ε, μεριά. Ε, θα πρέπει να δώσουμε μεγάλη μάχη ενάντια στην παράνομη διακίνηση και αυτό είναι το βασικό. Ε, τώρα έχουν επιστραφεί στην Τουρκία με βάση τη συμφωνία 1643 ε, και έχουν ε, ε, επιστραφεί με βάση τις εθελοντικές επιστροφές, δηλαδή το γεγονός ότι παίρνουν κάποια χρήματα και επιστρέφουν με τη δική τους θέληση, κοντά στα τελευταία δύο χρόνια, νομίζω ότι κοντά στα δύο μισή χρόνια, κοντά στις 20.000. και οι δύο οι τρόποι χρησιμοποιούνται, αλλά θέλω επειδή υπόθηκε μια ερώτηση να σας πω το εξής. Ε, οι διαδικασίες παροχής ασύλου πρέπει να είναι γρήγορες αλλά δεν μπορούν να είναι πρόχειρες. Υπάρχει και ένα δικαϊκό σύστημα και ένα σύστημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων που πρέπει να, ε, στο, το οποίο πρέπει να εκτελέσεις, πρέπει να το κάνεις. Τι κάνουμε λοιπόν εμείς, αυξάνουμε τον κόσμο που έχουμε για την εξέταση του ασύλου στα νησιά, καταγραφής και ασύλου. Ανέφερα ότι τους αυξάνουμε αυτό τον καιρό κατά 400 Αυξάνουμε τις επιτροπές προσφυγών από 12 σε 20. Εστιάζουμε αυτές τις 10 από αυτές τις 20 επιτροπές στα νησιά, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι, να ξεχνάμε για την δικό μας θέμα, ότι στην Ελλάδα συνολικά αυτή τη στιγμή βρίσκονται 568.000 μετανάστες από προηγούμενες περιόδους, πρώτης κρίσης δηλαδή του 2015. Ε, Αρκετοί από αυτούς είναι νόμιμοι, οι περισσότεροι είναι νόμιμοι, αλλά ο νόμιμος ο μετανάστης κάθε φορά χρειάζεται ανανέωση τα χαρτιά του, ε, κάποια στιγμή έχει χάσει τη, νομιμότητά του, χρειάζονται δηλαδή ε, τέτοια πράγματα. Αλλάξαμε ε, και τον τρόπο επίδοσης των αποφάσεων, αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο σε σχέση με την ταχύτητα. Ο δε στόχος μας είναι αυτή η διαδικασία, στόχος, στα νησιά να ολοκληρώνεται το πολύ σε 90 μέρες. Ώστε να ξέρει τώρα, εμείς αυτή τη στιγμή γνωρίζουμε ε, ότι υπάρχει μία διαδικασία η οποία λέει ε, της Ολλανδίας, μάλιστα έκανα και συνάντηση με τον ε, Ολλανδό Υπουργό, μια πολύ καλή συνάντηση για τον ευχαριστώ, ε, και μου είπε τη διαδικασία της ε, Ολλανδίας, δεν έχουμε την ίδια διαδικασία. Δηλαδή εμείς έχουμε ένα επίπεδο παραπάνω, αυτό συμβαίνει. Ε, εμείς θέλουμε να κατοχυρώσουμε όλα τα δικαιώματα, αλλά από την άλλη μεριά είναι και ένα θέμα, θα λέει, θα λέει κανένας, ποσότητας. Ποσότητας. Αν πάρουμε ε, τον τρόπο που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λέει να γίνει η κατανομή, με βάση το Δουβλίνο, η Ελλάδα θα πρέπει να εξετάζει περίπου 15.000 ε, αιτήματα ασύλου το χρόνο. Αυτή τη στιγμή εξετάζει 50.000 αιτήματα ασύλου το χρόνο. Και κάθε φορά όταν συζητάμε για αυτά χρειάζεται να συζητάμε και με ε, αριθμούς. Εμείς πάντως κοιτάμε τις πρακτικές κάθε κράτους ε, ώστε να προσπαθούμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί, αλλά σαφώς μόνιμα ε, δίκαιοι. Έρχομαι και τώρα στο, στο Δουβλίνο. Ε, καταρχήν, ε, μάλλον πριν από αυτό, μια απάντηση στο, στο ερώτημα του κυρίου ε, Χρυσόγονου. Όπως καταλαβαίνετε, και δεν μιλάω τώρα για την Ελλάδα, αν χώρες οι οποίες δέχονται προσφυγική πίεση, σε μια κατάσταση στασιμότητας και κλειστών συνόρων, χωρίς ανακατανομή, αρχίζουν και δέχονται και επιστροφές Βλήνου. και δεν σα λέω μόνο για την Ελλάδα, πάρτε την Ιταλία, πάρτε τη Μάλτα, την Κύπρο, την Ισπανία. Το θέμα θα γίνει πολύ μεγαλύτερο. Αν ας πούμε, ξέρω εγώ, έχουμε αυτή τη στιγμή, δεν είναι πάρα πολλέ, αλλά 500-600 αιτήματα του Βλήνου από τη Γερμανία, από την ε, Αλβανία σας είπα έχουμε τρία αλλά, που δεν είναι Δουβλίνου γιατί δεν συμμετέχει, αλλά είναι επανεισδοχή, αυτό το 500 θα προσθεθεί. Και εκεί που θα έχεις να κάνεις με, ας πούμε, πώς θα διαμορφώσεις την υποδοχή για 60.000 ανθρώπους, θα έχεις μετά, γιατί θα προσθεθεί και η Ολλανδία κτλ. Εμεί έχουμε πει, σε αυτή τη φάση που δεν υπάρχει το Δουβλίνο 4, να κάνουμε μία συζήτηση. Αλλά να το συνδέσουμε και με αυτό που λέει η κυρία Βόζεμπερκ το, το ζήτημα των επανενώσεων. Τυπικά δεν έχει παγώσει. Τυπικά δεν έχει παγώσει. Αλλά τώρα τι είναι αυτό που λέω κι εγώ. Τυπικά. Το θέμα είναι ότι πρακτικά δεν έχει γίνει μέσα στο 2018 καμία επανένωση που ήταν μια καλή πρακτική το προηγούμενο χρόνο. Και θα πρέπει εδώ να πω ότι η Γερμανία, για να, ε, τουλάχιστον η δικιά μου πλευρά του δίκαιου, έτσι το βλέπω, έχει προσφέρει πολλά στα ζητήματα της διαχείρισης του προσφυγικού μεταναστευτικού. Και θα πρέπει να στηριχθεί, γιατί στηρίζεται εν πολλής και το ολόκληρο το, το οικοδόμημα ε, σε αυτό που έχει κάνει ως τώρα και όχι να ανατρέψει αυτή την ε, λογική. Και πολύ περισσότερο κάτω από τη λογική ότι κάνουμε προετοιμασία μήπως ξανάρθει το 2015. Μα το 2015 δεν πρόκειται να ξανάρθει. Δεν υπάρχει ο πληθυσμό που θα... Λέω το λέω τελείω πρακτικά αυτό το πράγμα. Άρα νομίζω ότι εκεί πρέπει να μείνει. Ε, κλείνω με τα ζητήματα του, του Βλήνου. Κοιτάξτε, εγώ δεν θα ήμουν ε, τόσο εύκολος να πω ότι στις 28 του Ιουνίου δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Ε, ίσως αργότερα από ό,τι θα έπρεπε, αλλά βλέπω ότι έχουν κινητοποιηθεί όλοι σε αυτή την κατεύθυνση το τελευταίο χρονικό διάστημα, τις τελευταίες μέρες, είτε από το να μην υπάρχει, είτε από την πλευρά να υπάρχει. Και δεν συμφωνώ, δεν υπάρχουν απαντήσεις. Καταρχήν έχουμε μία απάντηση αυτή τη στιγμή και η οποία είναι και πάρα πολύ καλή πώς λύνεται το ζήτημα του Δουβλίνου και είναι η απάντηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δηλαδή η πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στην οποία καταλαβαίνετε και στα επιμέρους πολλές φορές αναφέρομαι, είναι μια πάρα πολύ καλή πρόταση. Αν με ρωτάτε, εγώ θα την ψήφιζα, δεν είμαι ευρωβουλευτή, θα την ψήφιζα με τα δύο χέρια. Αλλά συγχρονώ, όποιο έχει αντίθετη πρόταση, θα πρέπει να την πει. Ας πούμε, μια συμβιβαστική πρόταση στην οποία εμείς έχουμε δια... είναι της Βουλγαρικής Προεδρίας. Εμείς ας πούμε λέμε ότι πρέπει να είναι ο αναγκαστικός ο καταμερισμός και όχι εθελοντικός ο καταμερισμός. Λέμε ότι δεν μπορεί να υπάρχουν τόσες διαδικασίες και τόσες ψηφοφορίες. Λέμε ότι δεν, δεν πρέπει η πρώτη ευθύνη να πηγαίνει στα 8 χρόνια, αλλά μπορεί να πάει στα 2 ή στα 5. Σας λέω τώρα, είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε σε αυτό το πράγμα. Και συζητάμε σε αυτό το πράγμα. Υπάρχει όμως και η πλευρά η οποία λέει όλο αυτό απ' έξω. Φεύγει. Ε, λέμε ότι αυτό δεν είναι απάντηση. Αυτό δεν είναι απάντηση. Και δεν είναι δυνατόν μια ένωση που ξεκίνησε καταργώντας τα σύνορα να ορθώνει δύο ειδών σύνορα αυτή τη στιγμή το εξωτερικό της σύνορο και το εσωτερικό της σύνορο. Ή να το πω ας πούμε χαριτωμένα, σε μια δραματική κατάσταση χαριτωμένα, σκέφτομαι μερικές φορές, αυτοί οι άνθρωποι, οι πρόσφυγες, έρχονται προς την Ευρώπη ή εμείς ο δυτικός κόσμος τους στέλνουμε προς την Ευρώπη. Για σκεφτείτε το αν συνδράμουμε στους πολέμους που γίνεται στις περιοχές τους, ποιος στέλνει ποιον. Δηλαδή, δεν σας λέω, σας το, το λέω χαριτωμένο πρέπει να πάνω σε μια δραματική κατάσταση. Αλλά, για να το σκεφτούμε, μήπως αντί να συζητάμε αυτό, έπρεπε να συζητάμε πώς θα βοηθήσουμε τον Νίγηρα, πώς θα βοηθήσουμε την Ιγυρία, ώστε αυτοί οι άνθρωποι να μένουν στις πατρίδες τους, δεν θέλουν να φεύγουν, Πώς θα βοηθήσουμε ώστε να υπάρχει ειρήνευση στη Συρία, ειρήνευση στο Αφγανιστάν. Πώς θα, βοηθήσουμε ώστε να υπάρχει πυρηνική συμφωνία και όχι ο καθένας να τραβάει την υπογραφή του πίσω. Αλλά είμαστε πολλοί, με να το πω έτσι χοντρά και μην με θεωρήσετε ριζοσπάστη. Δεν είμαι. Είμαι αρκετά συμβαστικό άνθρωπος. Αλλά είμαστε πάρα πολύ καλά να ρίχνουμε τα σύνορα όταν συζητάμε για χρήματα. Είμαστε πάρα πολύ δεκτικοί και καλά κάνουμε στο να έχουμε ένα ενιαίο ευρωπαϊκό νόμισμα, να έχουμε μία ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα, αλλά ξαφνικά όταν ερχόμαστε στο ενιαίο σύστημα ασύλου, ο καθένας μιλάει για τη χώρα του. Ξαφνικά γίνεται ο καθένας για τη χώρα του. Σε αυτό επιτρέψτε μου να έχω διαφωνία ε, πλήρη. Ε, τώρα, αυτό είναι το ένα θέμα. Το δεύτερο θέμα, άρα εγώ θεωρώ ότι γίνονται προσπάθειες και μπορούμε να επιτύχουμε κάποιου του συμβιβασμό στις 28 του Ιούνιου, ώστε να αρχίσει το μεγάλο ζήτημα, η τρίλογη με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Για μένα είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό. Αν θέλετε την πρόβλεψή μου, αν δεν το πετύχουμε αυτό το πράγμα, τότε πάμε για να συζητάμε για το άσυλο μετά από χρόνια, όχι μετά από έξι μήνες που λένε μερικοί, ε, μετά από χρόνια. Δεύτερο ζήτημα, ανάφερα για τα ζητήματα της αλληλεγγύης, έχει μπει μια καινούργια ιδέα, η οποία όμως δεν έχει μπει επίσημα, την είδα τώρα τελευταία σε ένα χαρτί, νομίζω το πρώτο χαρτί, η οποία όμως δεν έχει αναλυθεί. Μιλάω για, αυτό, για, αυτή την περίφημη ιδέα περί εξωτερήκευσης των συνόρων, περί hot spot σε τρίτες ε, χώρες. Τι εννοούν με αυτή την ε, πρόταση. Και θέλω να θυμίσω ότι τέτοιες ενέργειες έχουν ξαναγίνει. Δεν θέλω να πάω πολύ πίσω στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά στη δεκαετία του 1990, σε σχέση με χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις χώρες του Μαγκρέμπ. Πού οδήγησαν όλα αυτά. Σε εντάσεις και δεν μπορώ να το πω διαφορετικά, και θανάτους αυτών ε, ανθρώπων, αλλά και σε εντάσεις μέσα στις ίδιες τις ε, χώρες. Δηλαδή είμαι πάρα πολύ φιδωλός, προσωπικά είμαι αντίθετος και προσωπικά διαβλέπω, και θα το κλείσω αυτό, μια προσπάθεια να αλλάξει η ατζέντα. Αντί να συζητάμε την αλληλεγγύη και την ανακατανομή, να συζητάμε τη θωράκιση και, να, να, συζητάμε το φόβο. Αυτό είναι το, το βασικό ζήτημα. Και ε, εγώ τώρα που έχω άποψη, την άποψη ότι η ασφάλεια είναι, προέρχεται από τη δημοκρατία, τι να πω σε σχέση με αυτό το πράγμα, όταν ο άλλος μου λέει η ασφάλεια είναι πάνω από τη δημοκρατία έχουμε μια διαφωνία <laughs> μερικές φορές. Φτάνει σε ένα επίπεδο που πλέον η συζήτηση δεν λέω ότι διακόπτεται, πάντοτε συνεχίζεται, αλλά φτάνει σε ένα ε, αδιέξοδο. Τελειώνω. Ε, κοιτάξτε, γνωρίζω τις ιδέες του κυρίου Πνάους. Ε, σας είπα για τις επιταχυντικές διαδικασίες που ε, εμείς ε, κάνουμε και τον παρακολουθώ πρέπει να σας πω ε, και το think ε, tank, όπως όμως παρακολουθώ και άλλα think tank. Δεν υπάρχει κάποιο think tank το οποίο έχει την αποκλειστικότητα, έχει την, ε, τουλάχιστον στη δική μου τη σκέψη. εγώ λέω ότι είναι βασικό ζήτημα η επιτάχυνση των διαδικασιών ασύλου. Είναι βασικό ζήτημα, αλλά αυτή η επιτάχυνση δεν μπορεί να γίνεται πρόχειρα, γιατί υπάρχουν και ορισμένες ιδέες μέσα σε αυτές τις ιδέες στις οποίες δεν θα συμφωνούσα. Σε καμία περίπτωση. Δηλαδή εγώ δεν μπορώ να βγω και να πω ότι οι Αφγανοί δεν δικαιούνται ε, εξέταση ασύλου. Ή δεν θα μπορούσα να πω ότι οι Σομαλοί, λέω αντίστοιχα, ή οι Νιγηριανοί δεν δικαιούνται εξέταση ασύλου. Ε, γι' αυτό σας λέω ότι είναι ένα ζήτημα προς, ε, όχι προ αλλά το παίρνω υπόψη μου, υπάρχουν ζητήματα που συμφωνώ. Τώρα για την ένταξη ε, είπα... Ε, μάλλον πριν από αυτό και για να τελειώσω, γιατί νομίζω ότι τελείωσε ο χρόνος μου και δεν θα το απαντήσω το άλλο. Ε, κοιτάξτε να δείτε τι, σκεφτόμαστε στο Υπουργείο. Αυτή τη στιγμή είναι 16.000 άνθρωποι στα ε, νησιά. Ε, υπολογίζουμε ότι κατά τη διάρκεια του Ιουλίου, του Αυγούστου και του Σεπτεμβρίου θα έρθουν στα νησιά περίπου τουλάχιστον άλλες 6.000 άνθρωποι. Οπότε δεν μετράμε με το 16.000, μετράμε με το 22.000. Και εμείς θέλουμε στο τέλος να έχουμε του Σεπτεμβρίου 10.000. Λέμε λοιπόν μέσα στον Ιούλιο οι ευάλωτοι να διαμορφώσουμε τέτοιες θέσεις στην υπηρετική Ελλάδα ώστε να απορροφήσουμε τους ευάλωτους. Ένας αριθμός τουλάχιστον 2.000. Να επιταχύνουμε τις διαδικασίες ασύλου και με ταχύ τρόπο να, να μεταφέρουμε... Τώρα εκεί μπαίνει και το ζήτημα των εθελοντικών και των με βάση τη δήλωση επιστροφών. Αλλά αυτό είναι ένα βασικό ζήτημα από τη μια μεριά πολιτικής, από την άλλη μεριά επιτάχυσης των διαδικασιών ασύλου. Θα τα κάνουμε και αυτά τα δύο και νομίζω ότι έχουμε όλη την καλή θέληση για να πετύχουμε. Μην ξεχνάμε όμως ότι το μεταναστευτικό προσφυγικό επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες. Ας πούμε η αύξηση των ροών το 2017-2018 κατά κύριο λόγο προήλθε από δύο γεγονότα. Το ένα γεγονός είναι ο πόλεμος στο Αφρίν. Το δεύτερο γεγονός μια γενικά μαζική έξοδο από το Ιράν και το Αφγανιστάν προς την Τουρκία. Άρα είχαμε μια ροή Κούρδων από την ε, μία μεριά, των ιτημένων δηλαδή, των ιτημένων στον πόλεμο εννοώ, ε, η οποία μας, ε, αν θέλετε, επηρεάζει. το ένα είναι αυτό και το δεύτερο είναι η μάχη με τους διακινητές. Και το τρίτο είναι πώς λύνουμε ζητήματα με την Τουρκία. Να το πω και αυτό και να το κλείσω. Η διαχείριση του μεταναστευτικού προσφυγικού από την πλευρά της Ευρώπης δεν μπορεί να γίνει αν δεν υπάρχει διάβλος επικοινωνίας και συζήτησης με την Τουρκία. Και όχι να κάνουμε τη συζήτηση επί ένα μήνα μετά τη συνάντηση της Βάρνας ποιος θα πληρώσει τα 3 δισεκατομμύρια πόσα θα πληρώσει ο ένας και πόσα θα πληρώσει ο άλλος και να γίνεται, ε, αν θέλετε, και στο τέλος ποιος, ποιος θα την πληρώνει η Ελλάδα, έτσι. <laughs> αυτό, αυτό, γίνεται. Γιατί ο άλλος χρησιμοποιεί δυστυχώ ανθρώπους, τους ανθρώπους, ως πίεση προς την Ευρώπη. Μα είναι δυνατόν. Όποιος με στρατιωτικούς όρους, το λέω αυτό γιατί ακούω κάτι για να βάλουμε στρατό στα σύνορα, όταν όποιος με στρατιωτικούς όρους πάει να λύσει ε, το προσφυγικό μεταναστευτικό, ε, από τη μια μεριά δεν θα το λύσει, από την άλλη μεριά θα τον εκδικηθεί η ιστορία. Σας ευχαριστώ πολύ. <clears throat> Ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ Δικαίω ε, σα χειροκρότησα να υπενθυμίσω ότι ήρθε χθε ο Υπουργό και απάντησε πολλέ λεπτομερεί ερωτήσει για την υπηρεσία ασύλου και η ομάδα του απαντούσε χθε. Οπότε η σχέση αυτή μεταξύ τη Επιτροπή μα ε, και του Υπουργού του Υπουργείου είναι πολύ ε, ισχυρή και για την ευρύτερη εικόνα εμείς δεν θα είμαστε στο Συμβούλιο, θα είναι ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, αλλά σωστά λέτε ότι η γραμμή της πλειοψηφίας εδώ μέσα είναι ξεκάθαρη. Εσείς ακούτε το τι θέλουν στο Συμβούλιο και βεβαίως και για το θέμα της εξωτερικής ανάθεσης δεν έχει δουλέψει ποτέ, δεν θα λειτουργήσει, μπορεί να είναι ελκυστική για κάποιους, αλλά δεν ε, θα λειτουργήσει. Θα είναι ένας εφιάλτης αν γίνει. Εμείς έχουμε μια πολιτική, είπαν κάποιοι συνάδελφοι, έχετε την στήριξή μας για να τα πείτε αυτά στις ε, συναντήσεις του Συμβουλίου. Και να τα έχουμε αυτά κατά νου και εδώ και στην ε, Ελλάδα. Σας ευχαριστούμε λοιπόν πάρα πολύ σήμερα και σας και την ομάδα σας κύριε Υπουργέ και καλή τύχη με τα όσα συμβαίνουν στα νησιά και στο Συμβούλιο. Σας ευχαριστούμε. Thank Σας ευχαριστώ και εγώ κύριε Πρόεδρε για την ε, φιλοξενία σας και την ευκαιρία που μου δώσατε να μιλήσω στους ευρωβουλευτές και ελπίζω να μην χάσατε το χρόνο σας ε, και ελπίζω να ανταλλάξουμε απόψεις ε, και πρακτικές ε, λύσεις σε κάθε θέμα και βεβαίως είστε πάντα ευπρόσδεκτοι αν θέλετε να έρθετε στην Ελλάδα να δείτε όχι μόνο εσείς, μια επιτροπή, κάποια αντιπροσωπεία, να δείτε οι ίδιοι το τι συμβαίνει στη Μόρια, στον Ελαιώνα, στη Ριτσόνα, σε όλα αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να αναφέρω πόσο οι συγητή για το Δουβλίνο και οι άλλοι συγητέ συνάδελφοι που έχουν επισκεφτεί τα νησιά είναι εδώ. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συνάδελφοι, περνάμε τώρα στο επόμενο θέμα, το οποίο είναι το σημείο 5, κατευθυντήριες γραμμές για τα κράτη-μέλη για να προληφθεί η ποινικοποίηση της ανθρωπιστικής βοήθειας. Εάν οι συνάδελφοι είναι έτοιμοι, μπορούμε να προχωρήσουμε. Οπότε, να σας εξηγήσω εδώ, συνάδελφοι, ε, για το ψήφισμα αυτό. Οι συντονιστές της ΛΥΜΠΕ αποφάσισαν στις 24 Μαΐου να υποβάλουν ένα ψήφισμα στην Ολομέλεια του Ιουλίου για να ζητήσουμε από την Κομισιόν κατευθυντήρες γραμμές για την εφαρμογή της λεγόμενης οδηγίας διευκόλυνσης. Η οδηγία αυτή ζητάει από τα κράτη-μέλη να εγκρίνουν τις ε, κατάλληλες ε, ποινές για άτομα τα οποία διευκολύνουν ε, παράνομη είσοδο και παραμονή. Προβλέπονται όμως εξαιρέσεις αν πρόκειται για ανθρωπιστικές περιπτώσεις. Οπότε ο στόχος θα είναι να υπάρξει μια σαφήνεια και ομοιόμορφη εφαρμογή με το να διευκρινίζει ποιες μορφές δεν θα πρέπει να ποινικοποιούνται από τα κράτη-μέλη. Εγώ, εισηγητής, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους και όδης εισηγητές για την γρήγορη δουλειά τους στο ευαίσθητο αυτό θέμα. Έχουμε ένα κείμενο το οποίο είναι στην διάθεσή σας σήμερα. Θα ψηφιστεί την Δευτέρα, 25 του μηνός. Το ψήφισμα έχει προετοιμαστεί κατόπιν τη συζήτηση και τη προφορική ερώτηση ε, στις 12 ε, Ιουνίου. Σύμφωνα με το άρθρο 128, τώρα θα ήθελα να δώσω τον λόγο κατευθείαν στους ε, σκιώδεις εισηγητές για να ακούσουμε την άποψή του. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να δώσω τον λόγο στον Φρανκ Έγγελ του ΕΛΚ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Κλοντ. αναφέρετε κι εσείς ότι με το ψήφισμα αυτό προσπαθούμε να ενισχύσουμε την ασφάλεια δικαίου, δικαίου όσον αφορά το τι ακριβώ συνιστά ε, την διευκόλυνση, την, ε, το ποινικό αδίκημα της ε, διευκόλυνσης κάποιου να περάσει παράνομα τα σύνορα. το οποίο πράγματι είναι κολάσιμο, αλλά έχουμε διαπιστώσει τα τελευταία χρόνια η ανθρωπιστική βοήθεια μπορεί να πέφτει θύμα διώξεων αυτούς που την παρέχει, ε, σαν να επρόκειτο για διακινητή. Και στο ψήφισμα αυτό ζητούμε να καταπτυσσούν κατευθυντήριες οδηγίες, έτσι ώστε να ξεκαθαρίζεται τι είδους βοήθεια μπορεί να θεωρηθεί νόμιμη και παραδεκτή, ανάλογα και με τις περιστάσεις. Θέλουμε να είναι ξεκάθαρο, και το αναφέρουμε στο ψήφισμα, ότι θα, πρέπει να προστατεύσουμε τις ανθρωπιστικές ε, οργανώσεις οι οποίες βοηθούν και οι οποίες συνεισφέρουν στην διάσωση Διευκρινίζουμε όμω επίση ότι και αυτέ οι πρωτοβουλίε θα πρέπει να γίνονται σε συντονισμό με τι επίσημε κρατικέ αρχέ. Δεν μπορούν να ε, εργάζονται εντελώ αυτόνομα έτσι ώστε να ξεκαθαριστεί τι συμβαίνει με αυτές τις ε, ανθρωπιστικές ε, οργανώσεις στη Μεσόγειο. Βεβαίω η κατάσταση και το γεωγραφική περιοχή για την οποία αναφερόμαστε δεν διευκολύνει καθόλου την κατάσταση. Για παράδειγμα, τα διεθνή ύδατα που βρίσκονται εκτό των χωρικών υδάτων της Λιβύης δημιουργούν μια δυσκολία. Ε, κανόνες όμως πρέπει να τους εφαρμόσουμε σε αυτήν την περιοχή του κόσμου, αυτή μα αφορά και θα πρέπει να είναι ξεκάθαρη για όλου. Σας ευχαριστούμε για αυτή την ε, επικοδομητική προσπάθεια που κάνετε. Αυτή η περιοχή είναι περίπλοκη και είναι σημαντικό η Επιτροπή μας να προσπαθήσει να βελτιώσει την ασφάλεια δικαίου για τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται στην περιοχή αυτή. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και θα περάσουμε στους ασκιώδες από την πλευρά του ECR. Κυρία Χαλάχο, δεν είναι... Κυρίως, συγγνώμη, Χαλάχο. Δεν είναι παρόν. Μήπως υπάρχει κάποιος άλλος εκπρόσωπος του ECR? Όχι. Η κυρία Βίκστρομ, ε, Σίλια Βίκστρομ είναι η σκιώδης του Εσάλντε. Δεν θέλετε το λόγο. Έχουμε κάποια προβλήματα με το μικρόφωνο μου. Το δικό μου μικρόφωνο δεν σβήνει, λέει ο πρόεδρος. Φανώ έχει υπάρξει κάποιο πρόβλημα με το σύστημα το, το ηχητικό τη αίθουσα. Ούτε οι διερμηνείς μπορούν να κλείσουν το μικρόφωνο του αυτή τη στιγμή. Θα πρέπει να αναζητήσουμε το τεχνικό. ρωτά ο πρόεδρος, για λόγου ταχύτητας, ε, μάλλον μήπως δουλεύει το δικό σας μικρόφωνο. Όχι, ε, ναι. θα γίνω σαν ηγέτης, ο ανώτατος ηγέτης η δικτατορία, μόνο το δικό μου μικρόφωνο θα είναι ανοιχτό, λέει ο πρόεδρος επόμενο.

συγγνώμη, λέει ο Πρόεδρος, θα πρέπει να κάνουμε ένα διάλειμμα 5 λεπτών για να επιληθεί το τεχνικό πρόβλημα με τα μικρόφωνα. Το λέω και για τους συναδέλφους που μόλις μπήκαν στην αίθουσα. Μόνο ένα μικρόφωνο λειτουργεί από τους ομιλητές, το, το μικρόφωνο του Προέδρου. Δυστυχώ και τα μικρόφωνα του διαμηνέων είναι όλα ανοιχτά. Θα βρούμε έναν τρόπο να το λύσουμε. οι τεχνικοί προσπαθούν να λύσουν το πρόβλημα. Θα σας ενημερώσω μόλι γνωρίζω τι, τι, έχει συμβεί. Θα χρειαστεί λίγο χρόνο ακόμα όμως. Λοιπόν, συνάδελφοι, θα το διαπιστώσατε κι εσείς, έχουμε ένα τεχνικό πρόβλημα. Δεν δουλεύει κανένα από τα μικρόφωνα στην αίθουσα των ομιλητών, μόνο το μικρόφωνο του Προέδρου. Αυτή τη στιγμή η τεχνική υπηρεσία προσπαθεί να το επιλύσει το πρόβλημα, αλλά δεν θα ήθελα να καθυστερήσουμε. Ε, με την άδεια σας θα ζητούσα να αρχίσουμε την ψηφοφορία. Αν κάποιος έχει αντίρρηση, παρακαλώ να μου το πει. Τώρα, αυτό σημαίνει ότι αν ε, θέλετε να πάρετε το λόγο κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας, σηκώστε το χέρι σας, θα μιλήσετε χωρίς μικροφόνου και θα δούμε τι θα γίνει με τη διερμηνία. Τώρα έχουμε πρόβλημα και τα μικροφόνα της διερμηνίας. Μπορούν να, να γίνει δεκτό αυτό. Άκουσαν όλοι αυτό που είπα. Ωραία. Θα προχωρήσω λοιπόν με την... Κύριε Μπέκα, σηκώνετε το χέρι για να πείτε ότι συμφωνείτε, ότι δεν έχετε πρόβλημα. Ωραία. Ε, θα προχωρήσουμε λοιπόν με την ψηφοφορία και δεν θα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα μικρόφωνα μέχρι να επιληθεί το τεχνικό πρόβλημα. Το προσπαθούν. Ωραία. Το πρώτο θέμα για την ψηφοφορία είναι το σημείο 6 προς σχέδιο, ε, σχέδιο έκθεση για τη χρήση του συστήματο πληροφοριών σύγκαινε για την επιστροφή των παρανόμω διαμένων των υπηκών τρίτων χωρών ε, για την α, Κροατία. Έχει ήδη διανεμηθεί σε το προσχέδιο του εισηγητή. Δεν θα του δώσω το λόγο, δεν θα ζητώσω το λόγο σε κανέναν γιατί δεν έχουμε τα μικρόφωνα και σα ζητώ κάτι εξαίρεση να το δεχτείτε αυτό στη διαδικασία. Εάν δεν υπάρχει εντήρηση λοιπόν προς αυτή τη διαδικασία θα έλεγα να προχωρήσουμε ε, με απλοποιημένη ψηφοφορία να εγκρίνουμε την ε, έκθεση. Σας ευχαριστώ. Πάμε τώρα στο επόμενο σημείο για την ψηφοφορία. Συγητής ο κ. Λενάχ για πρόταση κανονισμού του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σε σχέση με τη χρήση του συστήματο πληροφοριών Σέγγεν για την επιστροφή των παρανόμων διαμενών των υπηκών τρίτων χωρών, έναρξη ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορία. Εγκρίνεται με 39 ψήφους υπέρ και 7 κατά και δύο αποχές. Περνάμε στο επόμενο σημείο και πάλι κανονισμός Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου αφορά την εγκατάσταση, λειτουργία και χρήση του συστήματο πληροφοριών Σέγγεν. Ο εισηγητή ο κ. Κοέλιο. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρα τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Και πάλι έκθεση για το σύστημα Schengen, SIS του κ. Κοέλιο για ποινικέ υποθέσει. Έναρξη τη ψηφοφορία, παρακαλώ. Πέρα ψηφοφορία. Εγκρίνεται με 42 ψήφου υπέρ, 5 ε, κατά και μία αποχή. Α προχωρήσουμε στο επόμενο σημείο, προσχέδιο έκθεση για την έναρξη διαπραγματεύσεων για τη συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ιορδανίας σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τώρα, έχουμε μια σειρά εκθέσεων για οι, πολλές χώρες, η Ιορδανία, Τουρκία, υπάρχουν διάφορες τροπολογίε οι οποίε επαναλαμβάνονται. Στι περισσότερε περιπτώσει είχαμε καταφέρει να βρούμε ε, συμβιβαστικέ λύσει. Σα προτείνω λοιπόν το εξή. Να ξεκινήσουμε από το 2026, δηλαδή την Ιορδανία. Στον κατάλογο ψηφοφορία βλέπετε ποιε τροπολογίε ε, επαναλαμβάνονται. Θα θεωρήσουμε ότι αν εγκριθούν ή απορριφθούν στην ψηφοφορία για την Ιορδανία, εγκρίθηκαν ή απορρίφθηκαν αντιστοίχω και για τι υπόλοιπε εκθέσεις. Είναι ξεκάθαρη η διαδικασία. Είναι δύσκολα τα πράγματα σήμερα με το πρόβλημα με τα μικρόφωνα. Ε, πριν όλα πήγαιναν καλά, <laughs> πριν ξεκινήσουμε τη ψηφοφορία. τώρα ξαφνικά βλέπω ότι δεν υπάρχει διαφωνία με τη διαδικασία μου, και αλλιώς αν είπατε ότι διαφωνείτε δεν σας άκουσα. Ας προχωρήσουμε λοιπόν με την ψηφοφορία. Και Συνάδελφοι, σηκώστε το χέρι σας, εάν έχετε κάποια ένσταση επί της διαδικασίας. Ωραία. Σημείο 12, λοιπόν. Ένα της ψηφοφορίας. Πέρας ψηφοφορίας. Μάλιστα, απορρίπτεται. Ναι, ωραία, θα πηγαίνω πιο γρήγορα. 14 άρχεται η ψηφοφορία. 14. Πέρας. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 1. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. Συναδελφοί, έχω κάνει λάθος. Δεν ψηφίσαμε την 13. Ζητώ συγγνώμη. Να επανέλθουμε. Πάμε πίσω. Στην πρώτη σελίδα να ψηφίσουμε την 13. Άρχεται η ψηφοφορία. 13. Ψήφισαν όλοι πέρας. Δεκτή. Επιστρέφουμε λοιπόν. 19 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 2 αρχετή ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. Συμβιβαστική 3 αρχετή ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή συμβαστική 4 αρχετή ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. Συμβαστική 5. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. Συμβαστική 6. Άρχεται. Πέρας. Δεκτή. 33. Άρχεται. Πέρας. Δεκτή. 34. Άρχεται. Πέρας. Δεκτή. Α, απορρίπτεται, συγγνώμη. 36. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. Συμβιβαστική 7 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. 39 άρχεται η ψηφοφορία. Α, να ξαναγίνει. Ελπίζω να μην χαλάσει και το μηχάνημα της ψηφοφορίας. 39. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Μπορείτε να δοκιμάσετε κάποιο μικρόφωνο να δείτε αν δουλεύει. Απορρίπτεται. Ακόμα δεν δουλεύουν μάλιστα. 40. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Μάλιστα. 41. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. 42 αρχιετή ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. 43 αρχιετή ψηφοφορία. Πέρας. Απορριπτείται. 44 άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. 47 αρχιετή ψηφοφορία. Πέρας. Ψήφισαν όλοι. Ωραία. Απορρίπτεται. Τροπολογία 5 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Τοπολογία 5. 5. Ε, εξακολουθεί να είναι ανοιχτή η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. 6. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται η τροπολογία 7. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. 8. Αρχιτή ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. 9. Αρχιτή ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 10. Πέρας. Απορρίπτεται. Εκτιμώντας ε, τροπολογία 1. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή τροπολογία 2. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή τροπολογία 3. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Και τελική ψηφοφορία με ονομαστική ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Δεκτή. 44 υπέρ 2 ε, κατά 3 αποχές. Ωραία, συνάδελφοι. Τώρα περνάμε στην Τουρκία. Τροπολογία 14, αρχιετή ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 17, αρχιετή ψηφοφορία. Α, συγγνώμη. 17. Ψηφίζουμε ακόμα. Ακόμα στη 17 είμαστε. Η μηχανή είχε κολλήσει. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. 18 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Δεκτή. 19. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Δεκτή. 21. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρασε. Απορρίπτεται. 25. Άρχεται ψηφοφορία. Ναι, Τζούντιθ. Πρέπει να φωνάξεις. το είπα. Ε, είπα ότι φωνάζεις ούτω ή άλλω. Δυστυχώ δεν ακούμε. Λοιπόν, Τζοντίθ, ε, συγγνώμη που είπα ότι φωνάζει ούτω ή άλλω. και δεύτερον έχει δίκιο. Ναι, ναι, ναι. Συνάδελφοι, την προσοχή σα λίγο. Η κυρία Σαρτζεντίνη έχει δίκιο. Δεν ψηφίσαμε την τροπολογία 20. Και ευχαριστώ που το είδες. Δεν είναι τόσο δραματικά τα πράγματα. Ναι, δεν θα ξεκινήσουμε από την πρώτη μέρα τη δημιουργία. Λοιπόν, τροπολογία 20, άρχεται η ψηφοφορία. Ορίστε. Περιμένετε λίγο, για περιμένετε. Λοιπόν, Χριστίν, ακούστε και πείτε μου αν συμφωνείτε. Η 15 εγκρίνεται γιατί εγκρίθηκε στην Ιορδανία. Οπότε ίσως αυτό δεν έχει λάβει υπόψη. Και μετά έχουμε μόνο την τροπολογία 20 που πρέπει να ψηφιστεί, εντάξει. Οπότε επανερχόμαστε σε αυτό. Όχι, Είναι η τροπολογία 20 επί της παραγράφου 3. Πρέπει να ψηφίσουμε την 20, στην παράγραφο 3, τροπολογία 20. Όχι, όχι, δεν ισχύει αυτό που λέτε. Δεν θα καθυστερήσουμε άλλο. Λοιπόν, για να είμαι φύση 15 εγκρίθηκε, εγκρίθηκε στην ψηφοφορία για την Ιορδανία, οπότε έχουμε την 20. Αυτό ήταν το λάθος που είχε γίνει. Ναι, ναι, ναι, όχι, διάβασέ το. Λοιπόν, τροπολογία 20. Όχι, όχι, περνάμε στην 20. Ναι. Καταλαβαίνω τα όσα λέτε, αλλά πρέπει να ολοκληρωθεί ο κατάλογος ε, της ε, ψηφοφορίας. Λοιπόν, τροπολογία 20. Άρχεται η ψηφοφορία. Την 20 ψηφίζουμε. Ψήφισαν όλοι. Ακόμα και αν δεν θέλατε την 20. Πέρας. Απορρίπτεται. Οπότε τώρα περνάμε στην 25. Εντάξει. Τροπολογία 25, άρχεται η ψηφοφορία. Μάλιστα, 25. Πέρας. 25. Απορρίπτεται. 32. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Και απορρίπτεται. 36. αρχιετή ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Μάλιστα. 49 τώρα. στη σελίδα 8 του καταλόγου σας, 49. Ναι, εντάξει, μην λέω αριθμό σελίδα. Τροπολογία 49. Μπορείτε ακόμα να ψηφίσετε. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 51. Συγγνώμη, λάθος. Καταπίπτει. 60. Τροπολογία 60. Άρχεται η ψηφοφορία. Τροπολογία 60. Τι γίνεται. Ψήφισαν όλοι πέρας. Απορρίπτεται. Εκτιμώντας τροπολογία 5 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Και απορρίπτεται. Τροπολογία 6 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία άρχεται. Πέρας. Δεκτή. 49 υπέρ, 6 κατά. Και περνάμε γρήγορα στο Ισραήλ. Τροπολογία 14, άρχεται η ψηφοφορία. Στο Ισραήλ. Τροπολογία 14. Άρχεται η ψηφοφορία. Ανοιχτή είναι ακόμα η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλο το Ισραήλ. Κυρία Στίβενς, έχετε κάτι διαδικαστικό? Ωραία, να συνεχίσουμε να ψηφίσουμε. Περνάμε τώρα... Πέρασε η ψηφοφορία, συγγνώμη. Απορρίπτεται Τώρα μπορούμε να ψηφίσουμε την 18. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορία. Συμβαστική τροπολογία 1. Άρχεται η ψηφοφορία. Η προηγούμενη απορρίφθηκε. Πέραση ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Έχετε κάτι να, διαδικαστικό να πείτε, πέστε μου σας παρακαλώ. Και το μεταξύ είμαστε στην τροπολογία 11. Κυρία Στίβενς. Είμαστε στο Ισραήλ, δυστυχώς δεν ακούμε τα σχόλια της κυρίας Στίβης και είμαστε στην τροπολογία 11. Σας παρακαλώ, δείτε τον κατάλογο των ψηφοφοριών. Είμαστε στην ε, τροπολογία 11. Δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα, δεν θα επηρεάζονταν η ψηφοφορία. Τροπολογία 11, άρχεται η ψηφοφορία και είμαστε σίγουρα στο Ισραήλ. Σελίδα 9. Σελίδα 9 του καταλόγου ψηφοφοριών σας. Σελίδα 9. Παραμένει ανοιχτή η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Συγγνώμη, συγγνώμη. Ξέχασα την τροπολογία 43. Ούτε ξέρω τι κάνω σήμερα. Σελίδα 8, όχι σελίδα 9. Αντί για την 9 πηγαίνετε στην 8 και στη σελίδα 8 βρείτε τη την τροπολογία 43 και ψηφίζουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. 43 Ψήφισαν όλοι για τη 43, για τη σελίδα 8. Πέραση ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Τώρα πάμε στην 11. Αιτιολογικές σκέψεις. Άρχεται η ψηφοφορία, τροπολογία 11 σε αιτιολογικές σκέψεις. Πέραση ψηφοφορίας. εγκρίνεται και τώρα πάμε στην τροπολογία 4 τροπολογία 4 αιτιολογικές εκθέσεις Α, όχι, δεν ψηφίζουμε την τροπολογία 4. Πάμε στην τελική ψηφοφορία. Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Τελική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέραση ψηφοφορία. Εγκρίνεται 43 ψήφοι υπέρ, μία αποχή. Πάμε στην Τινησία τώρα. Τροπολογία 12 στην Τινησία. Άρχεται η ψηφοφορία, πέραση της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται και με χαρά να σας πω ότι ψηφίζουμε το τελικό κείμενο. Ένα δωράκι. Τελική ψηφοφορία για την Τινησία. Άρχεται η ψηφοφορία. Τελική ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε ψηφοφορία. Εκρίνεται. Πάμε στο Μαρόκο. Τροπολογία 12. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορία ψηφοφορίας. Απορρίπτεται και ψηφίζουμε το τελικό κείμενο. Με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορία. ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 41 ψήφοι υπέρ 2 κατά 5 εποχές Πάμε στο Λίβανο. Τροπολογία 12. Άρχεται η ψηφοφορία. Είμαστε στο Λίβανο. Ε, κάποιος λέει την Αίγυπτο για να με μπερδέψει, αλλά είμαστε στο Λίβανο. Οι σοσιαλιστές μπορούν να αποφασίσουν πώς θα ψηφίσουν. Παραμένει ανοιχτή η ψηφοφορία. Ωραία. Πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται. Τροπολογία 47 στη σελίδα 7 του καταλόγου σας. Τροπολογία 47, άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση τη ψηφοφορίας. Τελική ψηφοφορία απορρίπτεται και τώρα ε, ψηφίσουμε το τελικό κείμενο. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 42 ψήφοι υπέρ, 2 κατά, 5 εποχές. Τώρα πάμε στην Αίγυπτο. Τροπολογία 13. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Και πάμε στην τροπολογία 16. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 24. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται τροπολογία 25. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 42 στη σελίδα 7. Α, συγγνώμη μισό λεπτάκι. έχει καταπέσει 42 και πάμε στην 53 στη σελίδα 8. Τροπολογία 53, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας για την 53 απορρίπτεται στις αιτιολογικές σκέψεις τώρα τροπολογία 5 άρχεται η ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται Τελική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Και τώρα πάμε στην Αλγερία. Τροπολογία 12. Σαν παγκόσμιο πρωτάθλημα είναι. <laughs> Περίπου. τη ψηφοφορίας απορρίπτεται. Ψήφισες λάθος, Άννα. Πέραση ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Τροπολογία 47. Στη σελίδα 7. Τροπολογία 47. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Και πάμε στην τελική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορία. και εγκρίνεται. 41 ψήφοι υπέρ, 2 κατά, 5 αποχές. Τελείωσε λοιπόν η ψηφοφορία. Ευχαριστώ για την υπομονή σας συνάδελφοι. Συγγνώμη για τα λάθη. Συνάδελφοι, για το επόμενο σημείο οι τεχνικοί θα ξανακινήσουν το σύστημα για να λειτουργήσουν τα μικρόφωνα. Θα πρέπει να περιμένουμε λοιπόν τουλάχιστον 5 λεπτά. Διάλειμμα τουλάχιστον 5 λεπτών. Ευχαριστώ πολύ.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

Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ξεκινήσουμε με την ημερήσια διάταξη, θα συνεχίσουμε. Λειτουργούν τώρα τα μικρόφωνα. Ευχαριστούμε και τους τεχνικού που διόρθωσαν το πρόβλημα. Και πάμε στο σημείο 18. Αν είστε έτοιμοι. Είναι εδώ και ο κύριος ε, Μορντού, οπότε μπορούμε να ξεκινήσουμε. Sorry, colleagues, a very confusing morning. Συγγνώμη, συνάδελφοι, σήμερα το πρωινό είναι όλα ανάστατα. Δεν είχαμε τελειώσει το σημείο για τη διευκόλυνση και ξέρω ότι είναι τουλάχιστον ένα εκ των σκιωδών, η Μάλιν Πιόρ, και δυστυχώ ε, δεν μπορέσαμε να ακούσουμε την κυρία Βίξτρομ. Ο κύριος Έγκελ είχε μιλήσει, δεν ξέρω μήπως θα μπορούσαμε να τελειώσουμε με το σημείο αυτό, διότι θα ήταν ε, αδιανόητο να μην γίνει, σταμάτησαν να λειτουργούν τα μικρόφωνα εν μέσω της συζήτησης, αλλά έχουμε έναν εκ των σκιωδών. Μήπως θα μπορούσαμε να το συμπληρώσουμε το σημείο αυτό. Μάλιν. Ω και από πλευρά τη ΓΚΟΕ, θα μπορούσες να μας πεις την άποψή σου για το σχέδιο ψηφίσματος. Ευχαριστώ πολύ. Διευθυνή σήμερα πρεσφύγων σήμερα, επομένω είναι επίκαιρο και απαραίτητο αυτό το ψήφισμα και είναι πάρα πολύ σημαντικό. 27.000 θανάτους καταγράφουμε από πνιγμούς ε, στη Μεσόγειο και αυτή είναι η γνωστή θάνατη, επομένως ε, τα επίσημα στοιχεία μάλλον είναι υψηλότερα. Ε, εμείς πιστεύουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι ήρωες και σώζουν ζωές. Ε, τώρα, αν είναι σε αποστολές, σε μη κυβερνητικές οργανώσεις, σε ε, πολεμικά πλοία, εμπορικά πλοία, δεν έχει σημασία. Όποιος διασώζει ανθρώπινες ζωές στη θάλασσα είναι ήρωα. Η τελική κυβέρνηση που τώρα φαίνεται να ε, περηφανεύεται επειδή ε, παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και τις ανθρωπιστικές αρχές, είναι απλώς ένα βήμα ακόμα προς τον πάτο και εμείς πρέπει να κάνουμε κάτι για να το ανατρέψουμε αυτό. Πιστεύω ότι αν πραγματικά θέλουμε να έχουμε υψηλότερο ηθικό πλεονέκτημα από τον πρόεδρο των ΗΠΑ που τώρα χωρίζει οικογένειε ε, μητέρε από τα παιδιά του, πρέπει να τηρούμε και τι ανθρωπιστικέ αρχέ και τον νόμο. Η οδηγία για τη διευκόλυνση ήταν κάτι το οποίο επικρίναμε ευθύ εξ αρχή, αλλά υπάρχει αυτή η εξαίρεση ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να εξαιρούν την ανθρωπιστική βοήθεια. Επομένω, αν δεν υπάρχει κανένα οικονομικό όφελος, δεν θα πρέπει να τιμωρήσει. Γι' αυτό και θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα χρησιμοποιείται αυτή η εξαίρεση από τα κράτη-μέλη. Θέλουμε τις κατευθυντήριες γραμμές, αλλά θέλουμε να είναι απόλυτα σαφείς για το τι περιμένουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, Μάλιν. Ήταν ε, απογοητευτικό το γεγονός ότι διεκόπη το σημείο αυτό λόγω του τεχνικού προβλήματος. Η Τζούντιθ ε, Σαρχεντίνη ήταν εδώ και δεν είχε μιλήσει. Κάπου πετάχτηκε θα ξανάρθει. Δεν είμαι βέβαιος τι πρέπει να κάνω. Να πάμε απευθεία στο επόμενο σημείο. Εκτάκτος, όταν έρθει η κυρία Σαρχεντίνη θα της δώσουμε το λόγο για να πει δυο λόγια για το θέμα αυτό να πω ότι στη Λίμπη θα ψηφίσουμε στις 25 Ιουνίου για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ και πάλι για την υπομονή σας. Τώρα, πάμε στην ημερήσια διάταξη. Σημείο 18. Να καλωσορίσουμε τον κύριο Μόχτου. Έχουμε μια παρουσίαση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το πού βρίσκονται οι συμφωνίες επανεισδοχής ε, και άλλες ε, ευρωπαϊκές ρυθμίσεις ε, και το έργο της ε, κοινή Επιτροπής Επανεισδοχής ε, των κοινών μάλλον επιτροπών για την περίπτωση των συμφωνών επανεισδοχήν και να καλωσορίσουμε τον αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή, τον κύριο Μοχτή, και να ευχαριστήσω και τον Σάιμον, διότι πολύ συχνά έρχεται και μας ε, υποβάλει αναφορές εδώ. Το εκτιμούμε ιδιαίτερα ε, το γεγονός ότι έχει αναλάβει αυτή τη διέσμευση και είναι πολύ τακτικά εδώ. Η Κομισιόν βεβαίως έχει καθήκον να ενημερώνει τακτικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για όλες τις ε, συμφωνίες επανεισδοχής που συνάπτονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και επίσης κάθε έξι μήνες να ενημερώνει για την εφαρμογή αυτών των συμφωνιών και φυσικά το έργο των κοινών επιτροπών επανεισδοχή. Όπως ε, ζητήθηκε λοιπόν μα έδωσαν γραπτές πληροφορίες ε, για τι παρούσε συμφωνίε επανεισδοχή και άλλε ρυθμίσει που υπάρχουν και πριν δώσω το λόγο στον κύριο Μορτζή, θα ήθελα να τονίσω ότι από πλευράς Επιτροπής ΛΥΜΠΕ εξακολουθούμε να έχουμε ανησυχίε για την εξέλιξη αυτών των ε, ρυθμίσεων, οι οποίες μπορεί να παρακάμπτουν τις προτεραιότητές μας για τις διεθνείς συμφωνίες. Μια προειδοποίηση λοιπόν και πάλι για τις προτεραιότητές μας για το θέμα αυτό. Uh, Ευχαριστώ και πάλι λοιπόν που έρχεστε εδώ τακτικά να μας ε, ε, αναφέρετε τι συμβαίνει. Να σας δώσω το λόγο και ζητώ συγγνώμη για τις αποχωρήσεις μετά από την ψηφοφορία και όλα όσα συνέβησαν σήμερα το πρωί. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, από τα μέλη τη Επιτροπή Θεμελιωδών Ελευθεριών. Θέλω να σα ευχαριστήσω που μου δίνετε δυνατότητα να σα ενημερώσουμε και πάλι για τις δραστηριότητες μας, για το έργο μας, σε μία από τις πιο δύσκολες προκλήσεις που έχουμε στην διαχείριση της μετανάστευσης και είναι ακριβώς το ζήτημα το, της των, των προέλευσης και των επιστροφών. Στον αφορά τις επανεισδοχές, θα ήθελα να ξεκινήσουμε για να είναι ξεκάθαρο ότι δεν είναι η μόνη μας προτεραιότητα όσον αφορά τις προσπάθειες που κάνουμε στη διαχείριση της μετανάστευσης. Ουσιαστικός ο στόχος είναι να έχουμε ένα ε, σταθερό πλαίσιο που να βρίσκει μια σωστή ισορροπία ανάμεσα στην αλληλεγγύη και την ε, δικαιοσύνη. Ε, εδώ με τις επιστροφές προσπαθούμε να έχουμε μια ανθρώπινη αντιμετώπιση ενός φαινομένου που είναι ένα από τα πιο περίπλοκα και δύσκολα της εποχής μας. Προσπαθούμε δηλαδή να έχουμε ένα ουσιαστικό κοινό σύστημα ασύλου, να έχουμε νόμιμες διόδους προς την Ευρώπη και επίσης να συνεργαζόμαστε με χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσπαθώντας και να καταπολεμήσουμε τις γενεσιολογικές αιτίες της παράνομης μετανάστευσης και να προστατεύσουμε τους ε, παράτυπους μετανάστες αλλά και ε, επίσης να προστατεύσουμε τα εξωτερικά μας σύνορα. Υποστηρίζουμε διεθνείς οργανισμούς, τον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών, την Υπάτη Αρμοστία του για τους πρόσφυγες, τη Λιβύη, ε, στον Νίγηρα. Και για να σας δώσω ένα στατιστικό στοιχείο, από τότε που ξεκίνησε από το Μάιο του 2015 η πρωτοβουλία αυτή, είχαμε την δυνατότητα να βοηθήσουμε 25.000 μετανάστες και να τους βοηθήσουμε να τους επανεντεχθούν. Έχουμε επίσης ενισχύσει τις προσπάθειες μας να ε, καταπολεμήσουμε τη διακίνηση, τους διακινητές, ακριβώς εκείνους που ευθύνονται. Στον Ήγηρα το 2017 και μόνο είχαμε 26 συλλήψεις. 79 ε, διώξεις ασκήθηκαν για εμπορία ανθρώπων και επίσης ενισχύουμε τις προσπάθειες που κάνουμε για έρευνα και διάσωση στην έρημο, γιατί πολύ συχνά σκεφτόμαστε και ακούμε για την θάλασσα. Ε, μην ξεχνάμε ότι εκατοντάδες χιλιάδες, κατά δεκόσες ε, χιλιάδες άνθρωποι είχαν απλώς εγκαταληφθεί ε, στην έρημο από τους διακινητές τους. Αυτός... Έχουμε 140 προγράμματα πάνω από 4 δισεκατομμύρια ευρώ προπολογισμό. Σε μια δύσκολη συγκυρία προσπαθούμε να ενισχύσουμε, να ενθαρρύνουμε όλα τα κράτη-μέλη να ανοίξουν νόμιμε διόδου μετανάστευση και προγράμματα συνεργασία με τι αφρικανικέ χώρε. Ήθελα λοιπόν να ξεκινήσω από αυτά για να πω ότι έχουμε όλα αυτά τα μέτωπα ανοιχτά. Για να ε, ε, διευκρινίσω ότι δεν προσπαθούμε να χτίσουμε μια Ευρώπη φρούριο, αλλά μια Ευρώπη που θα είναι ανοιχτή σε αυτού που δικαιούνται προστασία αλλά για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε υψηλά πρότυπα ζωής, θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι πρέπει πρέπει να υπάρχει μια εξατομικευμένη διαδικασία ασύλου, η οποία να ξεχωρίζει εκείνου που δικαιούνται διεθνώ προστασία και εκείνου που δεν δικαιούνται. Και στη δεύτερη περίπτωση να υπάρχει μια διαδικασία για την επιστροφή του. Γνωρίζω ότι δεν έχουμε και πολλά, πολύ χρόνο στη διάθεσή μα, γιατί η διερμηνία θα είναι διαθέσιμη και μέχρι τι 12.30. Θα σα πρότεινα γι' αυτό το λόγο να μην σα διαβάσω πάλι ε, την επιστολή με τι πληροφορίε που σα έστειλα πριν από την συνάντησή μα, αλλά να σταθώ μόνο στι τελευταίε εξελίξει και ιδιαίτερα σε άλλες χώρες. Θα ήθελα να επαναλάβω η ευρωπαϊκή νομοθεσία εδώ είναι πολύ ξεκάθαρη. Η επιστροφή, η επέλαση δεν μπορεί να γίνει παρά μόνο μετά από εξατομικευμένη εξέταση της αιτησή του. Υπάρχει ασφαλιστική διεκλίδα για όλους τους ετούντε άσυλο που ζητάει από τα κράτη-μέλη να εξετάσουν κάθε υπόθεση ξεχωριστά για να αποφύγουμε την, την παραβίαση τη αρχής της μη επαναπροώθησης ε, ε, το είναι πολύ σημαντικό. Ε, αν λάβουμε υπόψη μας και το Μάιο, η Eurostat δημοσίευσε τα στοιχεία για τις επιστροφές του 2017. Είναι στην ιστοσελίδα από την προηγούμενη εβδομάδα. Φαίνεται ότι θα υπάρξει μια αύξηση των επιστροφών εξαιτία της μεγάλης εισρωής μεταναστών από το 2015 και 2016. Οι υποθέσεις οι οποίες περνούν από τη διαδικασία εξέτασης ασύλου και ταυτόχρονα υπάρχει και μια μείωση των ε, ποσοστών έχουμε φτάσει 31% στο ποσοστό ε, έγκριση των ετοιμάτων ασύλου του 2017 από πάνω από 40 που ήταν το 2015. Αυτό σημαίνει ότι και ο αριθμός εκείνων που θα επιστραφούν, που θα απελαθούν αυξάνεται. Ένα στοιχείο ενδιαφέρον είναι ότι από τα στοιχεία της Eurostat ότι παρά τη μεγάλη πολιτική ε, έμφαση που έχει δοθεί στο θέμα από... έχει μειωθεί ο αριθμός των επιστροφών από το 2006 μέχρι το 2017 το 2016 το 46% των απελάσεων εκτελέστηκαν, ενώ το 2017 το ποσοστό το αντίστοιχο είναι 36,6%. Για πολλούς λόγους, πιθανότατα ε, επειδή στο 2016 είχαμε μεγάλες επιστροφές από την περιοχή του Δυτικού Σουδάν ε, και οι προς χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, χώρες δηλαδή προς τις οποίες οι απελάσεις είναι ε, εφικτότερες, ευκολότερες. Η συνεργασία μας με διάφορες τρίτες χώρες λειτουργεί αποτελεσματικά κατά την άποψή μου κυρίως εξαιτία και των συμφωνιών επανεισδοχής και από την υποστήριξη που έχει παράσχει η Frontex. Αυτό σημαίνει ότι τα κράτη-μέλη όλο και περισσότερο μπορούν να εκτελέσουν τις αποφάσεις επιστροφής, τους απελάσεις τους και Διαπιστώνουμε όμως ότι ένας αριθμός μεταναστών από μη συνεργάσιμες χώρες, από χώρες δηλαδή οι οποίες δεν επιθυμούν να έχουν με εμάς συμφωνία επανεισδοχής, ο αριθμός αυτός αυξάνεται και αυτό σημαίνει ότι δημιουργείται ένα πρόβλημα γιατί όλο και περισσότεροι άνθρωποι βρίσκονται σε μια κατάσταση νομικής αβεβαιότητας, ανασφάλειας. Δεν έχουν ούτε δικαίωμα δομήμες παραμονή στην Ένωση, ούτε η χώρα τους τους δέχεται να γυρίσει πίσω. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να εντείνουμε την προσπάθεια μας συνεργασίας με τις τρίτες χώρες και επίσης να εντείνουμε τις προσπάθειες των κρατών μελών για τις, ε, την εκτέλεση των απελάσεων. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν να ενισχύσουμε την Ευρωπαϊκή Ακτοφυλακή. Η νέα της εντολή της δίνει τη δυνατότητα να ενισχύει και να ε, ε, υποστηρίζει τις εθνικές δραστηριότητες των κρατών μελών. Να σας δώσω ένα στοιχείο σχετικό. Φέτος μόνο οργάνωσε 111 επιχειρήσεις ε, ε, επιστροφών ε, στα κράτη-μέλη, ενώ το 2016 ο αντίστοιχο αριθμός ήταν 39. Βλέπετε δηλαδή μια σημαντική αύξηση. Ε, μόλις πρόσφατα μάλιστα συνήφθη μια σύμβαση που θα δώσει τη δυνατότητα να δημιουργηθεί ένα κονσόρσιο, ένα δίκτυο κρατών μελών. Από την 1η Ιουλίου θα ξεκινήσει την λειτουργία, ένα δίκτυο για τις απελάσεις που θα προσπαθήσει να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα αυτών των επιστροφών και προσπαθώντας επίσης να, εξετάσει την εθελοντική επιστροφή. Θα ήθελα να είμαι ξεκάθαρος ότι εμείς συνεχίσουμε να προτιμούμε και να προωθούμε την εθελοντική επιστροφή ως λύση. Ε, Φτάσαμε πια στο σημείο όλα τα κράτη-μέλη να έχουν ένα ε, σύστημα για τις εθελοντικές επιστροφές το οποίο να λειτουργεί. Σε πολλές περιπτώσεις για πολλά κράτη-μέλη η χρηματοδότηση έρχεται απευθείας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν δούμε τώρα τις εθελοντικές επιστροφές και εδώ διαπιστώνουμε μια μικρή μείωση ε, κατά 20% στα τελευταία στατιστικά στοιχεία. Όμως εδώ υπάρχει και μια σύνδεση ανάμεσα στις αναγκαστικές επιστροφές και τις εθελοντικές ε, επιστροφές. διαπιστώνουμε ότι η εθελοντική επιστροφή λειτουργεί όταν υπάρχει, επαπειλείται η απέλαση σε διαφορετική περίπτωση και γι' αυτόν τον λόγο ε, πρέπει να συνεχίσει να λειτουργεί το σύστημα των αναγκαστικών επιστροφών έτσι ώστε να είναι και κίνητρο για τις εθελοντικές. Χρειάζεται λοιπόν συνεργασία με τις ε, χώρες προέλευσης. Και εδώ πιστεύω ότι οι προσεγγίσεις, οι ευρωπαϊκές λύσεις μπορεί να λειτουργήσουν πολύ καλύτερα από τις διμερείς σχέσεις. Γιατί κάποια κράτη-μέλη έχουν τέτοιες διμερείς συμφωνίες, αλλά αυτό είναι εμβαλωματικό. Θα... Ε, έλεγα κύριε Πρόεδρε, γνωρίζω τη σημασία που αποδίδει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, στο να είναι αυτές οι συμφωνίες να παίρνουν νομικά δεσμευτική μορφή. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι το ίδιο επιθυμεί και η Επιτροπή. Ε, την επίσημη σύναψη μιας συμφωνίας επανεισδοχή δηλαδή. Ε, οποτεδήποτε αυτό είναι δυνατό και έχει συμβεί με τις περισσότερες χώρες, θα έλεγα με, τις, ε, με το μεγαλύτερο αριθμό του, τι περισσότερες. Αλλά θα πρέπει να γνωρίζει κανεί ότι ήδη στο διεθνές δίκαιο προβλέπεται η υποχρέωση μιας χώρας να αποδεχθεί την απέλαση του υπηκόου της που παράνομα βρίσκεται σε, άλλη χώρα και να αποδεχθεί να τον, την επιστροφή του σε αυτήν. Ε, γι' αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει να εστιάσει η συνεργασία μας στα αποτελέσματα με, ταυτόχρονη, ε, με ταυτόχρονα σεβασμό του διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου και για να συμβεί αυτό χρειάζονται και πρακτικές συμφωνίες ιδιαίτερα όταν έχουμε απέναντί μα συνομιλητέ οι οποίοι δεν επιθυμούν τη σύναψη μια νομικά δεσμευτική επίσημη συμφωνία επανεισδοχή. Επομένως έχουμε και αντίστοιχε τέτοιες διευθετήσει, οι οποίες δεν είναι νομικές ε, συμφωνίες, δεν ε, οδηγούν στη σύναψη μια νομικής συμφωνίας, αλλά είναι μια ε, πρακτική συμφωνία για το πώ λειτουργεί η απέλαση προς τη χώρα αυτή. Και θα έλεγα ότι κατά τη διάρκεια του 2017 αυτό λειτουργήσε. Μιας και μειώθηκε ο ρυθμός των αφήξεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξαιτία και των γενικότερων διεθνών προσπαθειών για να αντιθευτεί η μεταναστευτική κρίση βλέπουμε ότι αυτές οι συμφωνίες επανεσδοχής, αυτές οι νέες συμφωνίες έχουν αρχίσει να λειτουργούν αποτρεπτικά. Είναι δύσκολο να το αποδείξει κανείς αυτό με στατιστικά στοιχεία. Όμως βλέπουμε ότι και χώρες οι οποίες παραδοσιακά παλαιότερα όπως η Αιθιοπία, το Μπαγκλαντές, η Γουινέα ήταν μη συνεργάσιμες έχουν αρχίσει να αναλαμβάνουν τις ευθύνε τους, δηλαδή να αποδέχονται να γυρίσει σε αυτές ένας υπηκός τους από την Ευρωπαϊκή Ένωση με τα στο επίπεδο της πρακτικής διαδικασίας των ε, δικαιολογητικών. Ε, αυτό είναι μια σημαντική αλλαγή από την τελευταία φορά που ήρθα στην Επιτροπή σας να σας παράσχω μια ενημέρωση. Το διαπιστώνουμε ως τάση παρά το γεγονός ότι ε, τώρα σε αυτή την αρχική φάση ε, ο αριθμός των ανθρώπων που τους αφορά αυτή η κατάσταση είναι σχετικά μικρός. σε σχέση με τις προηγούμενες ενημερώσεις που σας έχω παρασχεί αυτή τη φορά σας έχω, έχω στείλει πολλά περισσότερα στατιστικά στοιχεία γι' αυτό πιστεύω δεν χρειάζεται να επαναλάβω τα γραπτά στοιχεία που σας είχαμε στείλει και ε, στην επιστολή μας στις 16 Μαΐου να σας ενημερώσω για εξελίξεις που έγιναν τους τελευταίους έξι μήνες. Να διευκρινίσω ότι το γεγονό ότι δεν θα αναφερθώ τώρα σε μια χώρα δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε στοιχεία. Θα μπορούσα να απαντήσω σχετικά στι ερωτήσει, στη διάρκεια των ερωτήσεων και των απαντήσεων. Ε, Του τελευταίου μήνε έχει ένα σημαντική πρόοδο. Γκάμπια. Εδώ δεν έχουμε νομικά δεσμευτική συμφωνία επανεσδοχή. Οι αρχέ τη Γκάμπια μα έχουν ενημερώσει ότι υπάρχει πολιτική συμφωνία από αυτού επί ενό κειμένου το οποίο περιγράφει τι βέλτιστε πρακτικέ για τι ε, διαδικασίε επανεσδοχή και το Μάιο ενημέρωσε και την πλευρά της Ευρωπαϊκή Ένωση ότι αποδέχεται το κείμενο αυτό. Επομένως θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται σε έξι μήνες από τώρα. Έχουμε τώρα κάνει τις απαραίτητες διευθετήσεις. Λοιπόν, για το Αφγανιστάν, μια πολύ ευαίσθητη χώρα, την οποία παρακολουθείτε πολύ στενά στο Κοινοβούλιο. Να ξεκινήσω με κάποια πολύ σημαντικά νέα, ότι δηλαδή στην τελευταία συνεδρίαση του Διαχειριστικού Συμβουλίου του ΕΑΖΟ τώρα υπό την Προεδρία μιας πολύ ικανής ε, εκτελεστικής διευθύντριας ε, ενέκρινε κατευθυντήριες γραμμές για το Αφγανιστάν. Δηλαδή προσπαθεί να κάνει μια κοινή αξιολόγηση για τις υπηρεσίες ασύλου των κρατομελών και μια ερμηνεία της κατάστασης που επίσης επιτρέπει για καλύτερη διάκριση μεταξύ διαφορών περιφερειών και περιοχών της χώρας. Ένα πάρα πολύ σημαντικό μέσο γιατί υποστηρίζει μια πολύ απαραίτητη σύγκληση των αποφάσεων περί ασύλου για το Αφγανιστάν. Το Αφγανιστάν εξακολουθεί να είναι μια πολύ σημαντική χώρα προέλευσης. Το 2016 ήταν η δεύτερη χώρα με πάνω από 180.000 ετούντες άσυλο. Έχει πέσει κάπως το 17 48.000 και είχαμε και σημαντική μείωση στο ποσοστό αναγνώρισης από το 60% στο 30% το 2017. Όπως γνωρίζετε υπογράψαμε την ε, συνεννόηση με το Αφγανιστάν το 2016, εφαρμόζεται νομίζω πάρα πολύ καλά και υπάρχουν και συμφωνίες επιστροφών και επανεισδοχής που λειτουργούν. Τον Μάιο στην Καμπούλ είχαμε την τέταρτη συνάντηση ομάδων εργασίας που περιέχουν και ζητήματα που αφορούν βίζες για συνοδούς ε, και το τι γίνεται για προξενικές υπηρεσίε εκεί όπου δεν υπάρχει αυγανική πρεσβεία. Γίνεται λοιπόν μια σαφής διάκριση ε, και κατά περίπτωση αξιολόγηση με τον Μπαγκλαντές ε, το 2017 η υπήκοοι Μπαγκλαντές ήταν η πρώτη υπηκοότητα μη Αφρικανών που έφταναν μέσω της κεντρικής Μεσογείου. Καταλήξαμε τώρα σε κάποιες τυποποιημένες διαδικασίες για την ταυτοποίηση και επιστροφή προσώπων που δεν έχουν άδεια παραμονής. Συμφωνήθηκαν αυτά πέρσι τον Σεπτέμβριο. Τον Απρίλιο είχαμε την δεύτερη κοινή ομάδα εργασίας όπου οι υπουργοί συμφώνησαν να προωθήσουν τις ε, περιπτώσεις εκείνες ε, όπου υπήρχε ταυτοποίηση αλλά δεν έχουν ακόμα να εκδοθεί ταξιδιωτικά έγγραφα και θα έλεγα ότι να επιβεβαιώνουμε την ε, στήριξη στην εφαρμογή αυτών των διαδικασιών. Τώρα η Αιθιοπία πάντα είναι ένα θέμα το οποίο σας ενδιαφέρει και σας ενδιαφέρει στο παρελθόν. Όπως γνωρίζετε συμφωνήσαμε σε διαδικασίες το 2017 για τις επιστροφές έχουμε ξεκάθαρες προθεσμίες και ορίστηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες για την έκδοση των ταξιδιωτικών εγγράφων. Αυτό είναι το βασικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε με πολλούς Αιθιώπες υπηκόους γιατί δεν υπάρχει δυνατότητα έκδοσης ταξιδιωτικών εγγράφων για μη εθελοντικέ επιστροφές ε, και τώρα έχουν αντιληφθεί ότι είναι μια διεθνή ε, υποχρέωση και πρέπει οι πρεσβείες τους να παρέχουν ταξιδιωτικά έγγραφα όταν βεβαιωθεί ότι είναι υπήκοοι και τέλος, ε, για να έχουμε και λίγο χρόνο στις ε, ερωτήσεις και απαντήσεις, η Γουινέα, η Γουινέα ήταν ε, πολύ ψηλά από τις τρεις κορυφαίες χώρες προέλευσης στην Κεντρική Μεσογειακή Οδό, αλλά συμφωνήσαμε με τις καλές πρακτικές τον Ιούλιο του 2017 και υπάρχει τώρα ένα πλαίσιο ταυτοποίησης επιστροφών κάτι το οποίο νομίζω τους ε, βοήθησε ιδιαίτερως γιατί έχουν προβλήματα διοικητικής ικανότητας οπότε βλέπουμε κάποια κράτη-μέλη αρχίζουν να χρησιμοποιούν τις διαδικασίες με θετικά αποτελέσματα αλλά εγώ θα ήθελα να δω τα κράτη-μέλη να χρησιμοποιήσουν περισσότερο την διαδικασία να αρχίσουμε να βλέπουμε και μια μικρή βελτίωση ε, των σχέσεων με τις προξενικές αρχές και τις πρώτες κοινέ επιχειρήσεις επιστροφών που γίνονται επιτυχώς Αργή πρόοδος λοιπόν, αλλά νομίζω ότι τώρα αρχίζουμε να βλέπουμε ε, την επιστροφή να γίνεται μια πιο ρεαλιστική προοπτική και επίσης και οι μη εθελοντικές επιστροφές ε, μας δίνουν την δυνατότητα να προωθήσουμε τις εθελοντικές επιστροφές με κάποια πακέτα ένταξης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λίγα λεπτά έχουμε. Λοιπόν, ε, κοιτάξτε, επειδή μετά τις 12.30 δεν θα υπάρχει πια διερμηνία, να ξεκινήσουμε με την Κριστίν. Μαρή Κριστίν, συγγνώμη. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Βερουζιά. Να σας υπενθυμίσω ότι σήμερα είναι η Διεθνή ημέρα Προσφύγων και ότι ο αριθμός των προσφύγων αυξήθηκε από πέρσι κατά 3 εκατομμύρια. Ότι τα 2 τρίτα των ε, ατόμων αυτών, ε, σύμφωνα με, τις, ε, με την ύπατη για τους πρόσφυγες, είναι από την Ιγυρία, από τη Σομαλία κλπ. Όταν σα ακούω, δεν είναι βέβαια η πρώτη φορά που ξέρω ότι υπάρχουν αυτέ οι συμφωνίες, δυσκολεύομαι να καταλάβω κάποια πράγματα. Καταρχά συμπεριφερόμαστε λε, και το καθεστώ ασύλου ήταν ομοιογενέ σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όλοι οι υπήκοοι τρίτων χωρών είχαν τι ίδιε δυνατότητε να λάβουν ε, άσυλο ανάλογα με τη χώρα. Ξέρουμε ότι δεν ισχύει αυτό. Δεν ισχύει, για παράδειγμα, για του Αφγανού. Υπάρχουν δευτερογενεί μετακινήσει όπω γνωρίζουμε, μεταξύ Γερμανία και Γαλλία, γιατί ε, η Γαλλία έχει βέβαια πολλά πράγματα στα οποία θα μπορούσαμε να την ε, επικρίνουμε, αλλά έχει υψηλότερο ε, ποσοστό ε, εγκρίσεων από τη Γερμανία. Σας ακούω να λέτε ότι προτιμάτε τις εθελοντικές επιτροπές με χαρά. Επιστροφές, συγγνώμη. νομίζω ότι εμείς θα πρέπει να δεχόμαστε μόνο αυτές και αυτό θα ήταν πιο σύνομο ε, κυρίως όσον αφορά την τρίτη χώρα και τα σχετικά άτομα. Λέτε ότι οι χώρε έχουν υποχρέωση να δεχτούν κάποιον ο οποίο έχει καταλήψει τη χώρα του. Ναι, αλλά υπάρχει και το άρθρο 13 τη Παγκόσμια Διακήρυξη των Δικαιωμάτων των Ανθρώπων. Λένε ότι ο καθένα έχει δικαίωμα να φύγει από τη χώρα του. Πώ μπορούμε λοιπόν να συμφιλιάσουμε τι δύο διεθνεί υποχρεώσει και κυρίω όταν ζητάμε από τι αρχέ, μάλλον λέμε ότι οι αρχέ πρέπει να δίνουν ταξιδιωτικά έγγραφα, ότι πρέπει να συμμετέχουν στη διαδικασία αναγνώρισης ταυτότητας. Ε, ανησυχώ ιδιαίτερα, για παράδειγμα, μας συζητούμε για την Αιθιοπία και ξέρω ότι ε, από τη ο Σουδάν ήρθαν κάποιοι, αναγνώρισαν κάποιους ε, Σουδανούς, επιστράφησαν κάποιοι από τη Γαλλία στο Σουδάν και αμέσως μόλις έφτασαν εκεί τους βασάνισαν. Ε, ξέρουμε λοιπόν ότι ξεφεύγουμε όλο και περισσότερα. Ε, λέμε ότι μειώνεται ο αριθμός των προσφύγων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ο αριθμό των ετούντων άσυλο μειώνεται, αλλά αν το συγκρίνουμε με αυτό το οποίο συμβαίνει στον κόσμο, πρόκειται για πραγματικό πρόβλημα και πρέπει να λάβουμε υπόψη και την παγκόσμια προσφυγική κρίση. Αλλιώ ε, ουσιαστικά κάνουμε ακριβώ το αντίθετο, την αγνοούμε. Ευχαριστώ, Ιάννα Γκόμε. Ευχαριστώ, κύριε Μορτού. Συμφωνώ σε κάθε λέξη με τα όσα είπε η συνάδελφος Μαρή Κριστίν Βερσιά. Και θα ήθελα να προσθέσω ότι μόλις επέστρεψε από μια αποστολή της Επιτροπής μας για την τρομοκρατία στην Κατάνια, όπου όντως επιβεβαιώσαμε ότι ο αριθμός των μεταναστών και προσφύγων που καταφθάνουν έχει μειωθεί ε, σε πολύ μεγάλο βαθμό μεν, αλλά ε, πλέον αντιλαμβάνομαι και επιβεβαίωσα εκεί ότι κάποια κράτη-μέλη δεν είναι απλώς ανίκανα και αδύναμα να κάνουν κάποια πράγματα, ε, αδιαφορούν για τις μαφίες της διακίνησης ανθρώπων που είναι αυτοί που διαχειρίζονται την ε, μεταφορά αυτών των ανθρώπων. Αν δω για παράδειγμα το ferry boat, το οποίο καθημερινά φέρνει ανθρώπους από τη Μάλτα στην Κατάνια ή ε, και στο που είδαμε το ferry boat και ξέρουμε, όπως γνωρίζουμε και εμείς, το γνωρίζει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο σκάνδαλο για ε, προγράμματα ε, ε, προστασίας για να πουλήσουν ε, ε ταυτότητες και διαβατήρια σε υπηκόους από, το από την Αλγερία κατά χιλιάδες παίρνουν θεώρηση από τη Μάλτα και όποιο πάρει θεώρηση μετά μπαίνουν σε ένα ferry και δεν υπάρχει κανένα έλεγχο στην Κατάνια, όπω μα είπαν οι ίδιε οι Ιταλικέ αρχέ. Τουλάχιστον όχι στου λιμάνες, ε, στους λιμένες. Ε, έχουν υπάρξει προβλήματα, υποτίθεται, στο αεροδρόμιο, ακριβώ ε, με τι ίδιε παράνομε θεωρήσει διαβατηρίων. Κάποιες χώρες λοιπόν Θέλουν απλώς να διαχειρίζονται τις ροές οι διακινητές. Και αυτό θα ήθελα να σας το ρωτήσω γιατί το αναφέρατε κι εσείς. Είπατε ότι υπάρχει ένα πρόγραμμα το οποίο υποστηρίζει η Πατέρμοστία, ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης κλπ. για επιστροφές ε, ε, από τη Λιβύη, προσφύγων από τη Λιβύη στις χώρες τους. Τι έχει να πει η Επιτροπή για το γεγονός ότι ο πρόσφατος κατάλογος κυρώσεων στη Λιβύη περιλαμβάνει και έξι ανθρώπους, τρεις εκ των οποίων ήταν ε, επικεφαλής παραστρατιωτικών οργανώσεων και ε, τρεις ε, από αυτές είναι γνωστό ότι χρηματοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και διοικούν τα κέντρα κράτησης, στα οποία έχουν βασανισμούς και άλλες κακοποίησεις και ε, ουσιαστικά διαχειρίζονται και τα δίκτυα που βάζουν αυτούς τους ανθρώπους στα σκάφη, στα πλοία, για παράδειγμα της επιχείρησης Σοφία ε, τα πλοία δεν μπορούν να πάνε να κάνουν διάσωση. Υπάρχει ο φασιστή ο Σαλβίνη, ο οποίο κατηγορεί τι μη κυβερνητικέ οργανώσει, αλλά οι μη κυβερνητικέ οργανώσει διασώζουν αυτού του ανθρώπου γιατί αλλιώ δεν θα του σώσει κανεί. Ε, η δική μας η αποστολή της ΚΕΠΑ, η CUNA4MED, δεν έχει εντολή να διασώσει ανθρώπους. Βεβαίως, εάν τους βρουν κατά μεσής της θάλασσας σε διεθνή δεν θα τους διασώσουν, αλλά δεν έχουν εντολή να πάνε να τους διασώσουν. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να πάνε οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις να κάνουν τη διάσωση. Και η ερώτησή μου προ εσά, κύριε Μορτού, και το αναφέρετε αυτό το πρόγραμμα, είναι μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας πει τι γίνεται με τα χρήματα τα οποία εκταμιεύονται για τη χρηματοδότηση αυτών των ανθρώπων που γνωρίζουν, που είναι γνωστοί και είναι στον κατάλογο των κυρώσεων των Ηνωμένων Εθνών. Πώς μπορεί να συνεχίζεται αυτή την κατάσταση, Πώ μπορούν τα κράτη μα να μην αναλαμβάνουν τι ευθύνε τη, του κατηγορώ διότι ε, εν γνώση Ε, διευκολύνουν αυτούς τους διακινητές ε, οι οποίοι διαχειρίζονται τη μεταφορά ανθρώπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι διερμηνείς θα σταματήσουν αυστηρά στις 12.30 λόγω των ε, κινητοποίησεών τους. Να πω, Τζούντιθ, ότι τελειώσαμε με το θέμα της διευκόλυσης, αλλά αν θέλεις να στείλεις κάτι γραπτός, ε, πολύ ευχαριστώ. Και είσαι και η τελευταία που θα λάβεις το λόγο και μετά θα πάρει το λόγο ο κ. Μορτού. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Υποστηρίζω τις κινητοποίησεις των διερμηνέων. Κυρία Μαχτού, σας ευχαριστούμε για την επιστολή και σας ε, ευχαριστούμε για το γεγονός ότι η ενημέρωση που μας παρέχετε γίνεται σε αιτήσια βάση. Πια αυτό είναι εξαιρετικό. Βέβαια, πάντα κάτι περισσότερο μπορεί να ζητήσει κανείς. Την επόμενη φορά, όταν αναφέρεστε ε, γραπτά σε κάποιες χώρες. Μήπως θα μπορούσαμε να είχαμε και κάποιο, ε, κάποια αριθμητικά στοιχεία σε ένα πίνακα. Αναφερθήκατε στην Αιθιοπία ε, και φαντάζομαι ότι ο αριθμός των επιστροφών θα είναι μικρός. Αλλά θα ήταν χρήσιμο να έχουμε αριθμητικά στοιχεία για όλε τι χώρε, όχι μόνο αυτέ που είναι υψηλά, αλλά και χαμηλά στον αριθμό των επιστροφών, για να έχουμε μια συνολική εικόνα το πώ λειτουργούν όλε οι συμφωνίε επανεισδοχή, είτε οι επίσημε είτε οι ανεπίσημε που περιγράψατε. Τώρα, ε, δεν σας άκουσα από την αρχή, ίσως το καλύψατε, ζητώ συγγνώμη τότε. Μπορείτε όμως να μου πείτε, στις διαπραγματεύσεις με την Τινησία και το Μαρόκο, ε, ένα από τα προβλήματα είναι ότι η, Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ζητάει μόνο οι χώρες αυτές να αποδέχονται την επιστροφή των υπηκόων τους, αλλά επίσης και όλων όσοι μπορεί να έχουν ταξιδέψει μέσα από την, την Ισία και το Μαρόκο και ε, δικαιολογημένα πιστεύω αυτές οι χώρες ε, εξανίστανται σε αυτό. Πώς μπορούμε να προωθήσουμε τέτοιες συμφωνίες γιατί κατά την άποψή μου και παράλληλα τις επικρίσεις για να έχουμε πολιτική ασύλου χρειαζόμαστε και πολιτική επιστροφών. Θα ήθελα να με ενημερώσετε λοιπόν τι έχει γίνει σχετικά. Ε, έχει υπάρξει πρόοδο, εάν όχι, μήπω κάνουμε κάτι για να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε τέτοια πρόοδο. Τώρα για την οποία διαπιστώνω ότι είναι και στην ευριανή μα ημερήσια διάταξη. Είναι καλό αυτό γιατί πράγματι πιστεύω ότι τα ερωτήματα αυτά θα πρέπει να τεθούν όποτε τη σωστή στιγμή, αλλά θα το προσπαθήσω και τώρα. Το οικοδόμημα αυτό είναι περίπλοκο. Είναι μια συμφωνία η οποία δεν έχει δημοσιοποιηθεί, αλλά διέρευσε στον τύπο. Ήταν μια συμφωνία η οποία εγκρίθηκε από σύνθεση του Συμβουλίου, άσχετη εμποροκυπένο ήταν η Υπουργή ε, Γεωργίας, δεν έχει σημασία. Ε, λέγεται ότι δεν δημιουργεί ε, δικαιώματα αλλά επίσης διευκρινίζει ότι μιλούμε ότι η Αιθιοπία δέχεται και θελοντικές επιστροφές αλλά και μη θελοντικές επιστροφές. Αυτό πιστεύω ότι έρχεται σε αντίθεση με την προσπάθεια που είχαμε κάνει με τις, να έχουμε μια σχέση με τις αφρικανικές χώρες που να βασίζεται στις εθελοντικές επιστροφές και ούτε με αυτά που μα λέει το Αμπιτζάν ότι εκείνοι θα δέχονται μόνο εθελοντικέ επιστροφέ. Μπορείτε να μου διευκρινίσετε τι γίνεται εδώ. Τι είναι αυτό το κείμενο που δεν είναι νομοθεσία, που, δεν έχει, που έχει κάπως εγκριθεί στο Συμβούλιο. πώ ε, θα χρησιμοποιηθεί αυτό ως βάση για την επιστροφή ανθρώπων και παρεπιπτόντως πότε θα το δει αυτό το κείμενο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. κύριος Μοχντού θα έχει δύο λεπτά στη διάθεσή του για να απαντήσει με διερμηνία. Μετά θα συνεχίσουμε μονάχα στα αγγλικά, λέει ο πρόεδρος. πρόεδρος ο κύριος Μοχντού. Θα ξεκινήσω απαντώντας στην κυρία Βίσια. Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι καμία μη εθελοντική επιστροφή, απέλαση δηλαδή, δεν είναι εφικτή εάν δεν έχει ακολουθηθεί προηγουμένως μια εξετομικευμένη εξέταση της αίτηση ασύλου. Εξετομικευμένη σημαίνει ότι θα πρέπει να δει την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα στην οποία, από την οποία προέρχεται τον άσυλο και επίσης πρέπει να προβλέπει διαδικασίες προσφυγής και δικαστικές, έτσι ώστε αν διαφωνεί ο άσυλο να μπορεί να προσφύγει σε ένα δικαστήριο κατά τις απόφασεις του. Ποτέ δεν συζητούμε για επαναπροώθηση ατόμων προς τα οποία έχει χορηγηθεί άσυλο. Μιλούμε μόνο για την απέλαση εκείνων που μετά την εξέταση του αιτήματο ασύλου του η διαδικασία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι αυτή η αίτηση ασύλου δεν είχε βάση. Βεβαίως, έχετε δίκιο που επισημαίνεται ότι υπάρχουν σημαντικές ε, διαφορές μεταξύ των ποσοστών αναγνώρισης από κράτος μέλος σε κράτος μέλος. Εσείς, αν δεν κάνω αναφερθήκατε στο ποσοστό αναγνώρισης του τον άσυλο από το Αφγανιστάν. Έχουμε από 1% σε κάποια χώρα και 19% σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και το συμπέρασμα το πολιτικό που εγώ ξάγω από αυτό είναι ότι γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό που η ΆΣΟ καταλήγει σε αυτές τις κατευθυντήριες οδηγίες για τις χώρες πρώτης εισόδου έτσι ώστε να υπάρχει μια βασική κατανόηση ε, της κατάστασης που επικρατεί σε κάθε μια από τις τρίτες χώρες έτσι ώστε να υπάρξει μια κάποια σύγκληση των αποφάσεων ασύλου στα κράτη-μέλη και πιστεύω ότι είναι σημαντικό αυτή, ε, σημαντική αυτή η προσπάθεια που γίνεται η Άσο να, να μετατραπεί σε υπηρεσία, ευρωπαϊκή υπηρεσία για το άσυλο που να δώσει μεγαλύτερη συνεκτικότητα στον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται η πολιτική ασύλου σε όλη την Ένωση και να αποτρέψει εκείνους που θέλουν να επιλέξουν τη χώρα στην οποία θα ε, υποβάλλουν το αίτημά τους. Επαναλαμβάνω ότι εμάς η πολιτική μας προτεραιότητα και προτίμηση είναι προς τις εθελοντικές επιστροφές. Όμως, όπως έλεγα, η εθελοντική επιστροφή γίνεται αποδεκτή από εκείνους ε, που ε, μπορεί να την ε, δεχτούν μόνο όταν γνωρίζουν ότι επαπειλείται σε, άλλη περίπτωση, σε διαφορετική περίπτωση η μη εθελοντική τους επιστροφή, η απέλασή τους. Έτσι έχουν τα πράγματα σε αυτό το τομέα. Επίσης, οποτεδήποτε οργανώνουμε μια επιχείρηση επιστροφής ή οποτεδήποτε καταλήγει σε ένα συμπέρασμα διαδικασία έλου, ο σεβασμό τη αρχή του νόχου εφουλμών τη μη επαναπροώθηση είναι αδιαπραγμάτευτο. Κύριε Γκόμε, αναφερθήκατε στα έξι πρόσωπα εναντίον των οποίων το Συμβούλιο Ασφαλεία του ΟΗΕ ενέκρινε κυρώσει. θα επικοινωνήσω με τους συναδέλφους που έχουν ασχοληθεί με το θέμα της παροχής τεχνικής βοήθειας προς την Λιβική ακτοφυλακή για να διευκρινίσω εάν έχει λάβει ευρωπαϊκή χρηματοδότηση κανένας από αυτούς. Οι διερμηνείς θα διακόψουν εδώ την παροχή της διερμηνίας. Mr. Milad from the Zawiya uh, Coast Guard, Libyan, so-called Libyan Coast Guard unit in Zawiya.